Καλημέρα σας. Έχουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία στι 9.30 και πρώτη συζήτηση είναι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2010 και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην εισηγητρία την κυρία Χίρης. Παρακαλώ. Ähm, äh, äh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι επιτροπή γυναικών και ίσων ευκαιριών. Εμείς γνωμοδοτούμε. Προσπάθησα τουλάχιστον να αναφέρω τα σημαντικά ζητήματα στη γνωμοδότησή μου και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και θετικές εξελίξεις αλλά Τώρα, σε εποχές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, συχνά ε, εκμεταλλεύεται ο κόσμος στο ε, επιχείρημα αυτό για να ασκήσει κακή πολιτική. Παρά τις εποχές της κρίσης, ε, λοιπόν, ε, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ε, η πολιτική ισότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα και ουσιαστικά είναι κάτι αυτονόητο. Το δεύτερο ε, θέμα είναι ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ε, ζωής. Ε, πολύ μας ενδιαφέρει η φροντίδα των παιδιών. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν επενδύσεις στην φροντίδα των παιδιών και να την αναπτύξουν. Επίσης, Επίσης η φροντίδα στο σπίτι γίνεται συνήθως από γυναίκες και μάλιστα συχνά θελοντικά. Ε, όταν ε, μέλη της οικογένειας, που συνήθως είναι οι κόρες, ε, δηλώνουν διατεθειμένες να φροντίσουν κάποια άλλη μέλη της οικογένειας, θα πρέπει και εδώ να βρεθεί μια φόρμουλα. Ε, έχουμε δηλαδή από τη μία την φροντίδα των παιδιών, από την άλλη έχουμε την φροντίδα κυρίως των γονέων, γενικά των ηλικιωμένων. Συχνά συζητάμε την ε, προσέλκυση εργατικού δυναμικού ε, από τις τρίτες χώρες, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο δυναμικό στις γυναίκες που πολύ συχνά είναι ειδικευμένε σε υψηλό βαθμό. Πολύ ε, σημαντική πρόκληση λοιπόν είναι να εκμεταλλευτούμε και αυτό το δυναμικό. Παρότι οι γυναίκες είναι ειδικευμένες σε μεγάλο βαθμό, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά τους μισθούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξή μας Ε, επίσης υπάρχει και μεγαλύτερος κίνδυνος απόλυσης ε, των γυναικών, ιδιαίτερα ε, σε μεγάλες ηλικίες. Κάτι άλλο που παίζει σημαντικό ρόλο είναι ότι νέα κορίτσια θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να μην επιλέγουν γυναικείες εντό εισαγωγικών δουλειές θα είναι ενδιαφέρον να ε, εξετάσουν ε, την ε, δυνατότητα να γίνουν μηχανικοί, να εργαστούν στις οικοδομές και τέτοια. Γενικά θεωρείται ότι οι γυναίκες γενετικά είναι κατάλληλες για κάποιες δουλειές, αλλά καλό θα είναι να μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα, να έχουν την επιλογή να κάνουν και άλλα επαγγέλματα. Επίσης, όσον αφορά τις μετανάστριες, ε, συζητάμε πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν, ε, αυτά που τους προσφέρονται. Γυναίκες που προέρχονται από άλλες ε, χώρες, ε, εάν έχουν ε, δικό τους επάγγελμα, αν κάνουν κάποια δουλειά, μπορούν να γίνουν πιο ανεξάρτητες. Το άλλο σημαντικό θέμα είναι το gender budgeting, το, η συμπερίληψη της διάστασης το, της των φύλων στον προϋπολογισμό. Σημαντικό είναι να υπάρχει συνείδηση πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ένα πολύ ωραίο και κλασικό παράδειγμα είναι σε σε δημοτικό επίπεδο η προώθηση του αθλητισμού. Ε, συχνά οι πόροι που υπάρχουν χρησιμοποιούνται για το ποδόσφαιρο, το οποίο μας αφορά κυρίως τους άντρες. Και τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ε, σε πράγματα από τα οποία να μπορούν να αποφεληθούν, διότι κανείς δεν σκέφτεται τη διάσταση αυτή. Επίσης, ε, Όσον αφορά ε, άλλους τομείς του προϋπολογισμού, σημαντικό είναι να ε, σκεφτούν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, τα χρήματα να πηγαίνουν κάπου όπου να μπορούν να επωφεληθούν και άντρες και γυναίκες. Επίσης έχουμε τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, ιδιαίτερα σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Ε, είναι πολύ ε, χρήσιμο να υπάρχει μια ποσόστοση ε, που να αντιστοιχεί ε, στη, στο ποσοστό των γυναικών ε, στο εργατικό δυναμικό συναλλικά. Εννοείται ότι εάν ε, μια επιχείρηση έχει μόνο άντρες εργαζομένους δεν έχει νόημα να, είναι γυναίκα, να υπάρχει γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο. υπάρχουν όμως για παράδειγμα πανεπιστήμια όπου όλες οι φοιτήτριες είναι κοπέλες και, ενώ όλοι οι καθηγητές είναι άντρες. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες ε, προτάσεις ε, και προσλέπω στην καλή συζήτηση και ε, στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στέινερ, και κατόπιν κυρία Λόπες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Χίρς για την έκθεσή της και σε κάποια σημεία μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία, πιστεύω. Η ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια και ε, εν μέρη οι εξελίξεις προχωράνε με ρυθμό χελώνας. Θα πρέπει να σκεφτούμε με ε, διαφορετικό τρόπο, να δούμε πού οι πρωτοβουλίες μας έχουν επιφέρει αλλαγές. η καινοτόμα σκέψη είναι απαραίτητη και εντός των επιχειρήσεων και όσον αφορά τις συνθήκες πλαίσιο για τις γυναίκες. Ε, και σε επίπεδο κοινωνίας όμως θα πρέπει να ε, σκεφτούμε διαφορετικά και όσον αφορά το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ε, ζωής, την φροντίδα των παιδιών. Στην ε, η Γερμανία υπάρχει η έκφραση ε, η, γυναίκα κοράκι που εγκαταλείπει τα παιδιά της δηλαδή και ε, αυτό πολύ συχνά αποθαρρύνει τις γυναίκες να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία. Εάν η άνδρες ε, συμμετέχουν εξίσου στην ε, ανατροφή των παιδιών, ε, τότε και ο εργοδότης ποτέ δεν θα ξέρει ποιος θα κάνει πιο, πιο πολλές απουσίες, ο, ο άντρας ή η γυναίκα εργαζόμενη. Και έτσι θα εξαλειφθούν πολλές από τις διακρίσεις βάρος των γυναικών. Επίσης, πολύ λίγες, έχουν, πολύ λίγες γυναίκες έχουν ε, χρόνο για εθελοντική εργασία. Δεν συμφωνώ απόλυτα στο θέμα αυτό με την κυρία Χίρς. Όσον αφορά τα σχέδια περί ισότητας ε, στην Ισπανία, υπάρχει ένα υποχρεωτικό σχέδιο ισότητας στο οποίο συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το επιδιώξουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το gender budgeting, είναι κάτι το οποίο εν μέρει εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Ε, είναι ένας δρόμος τον οποίο καλύπτουμε βήμα-βήμα, αλλά είναι μια διάσταση η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί στα κράτη-μέλη. Ε, πάντως προσβλέπω και εγώ στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λόπες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λόπε Φοντάνη. Ε, σας ευχαριστώ. Όπως ε, και η έκθεση της δικής μας αλλά και η έκθεση και επί της ουσίας, ε, είναι πολύ ορθά κείμενα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλό το κείμενο της συναδελφούς και είμαι ότι θα συμφωνήσουμε σε ένα συνενετικό κείμενο. Θα ήθελα μόνο να πω το εξή: Εγώ πιστεύω ότι είναι κρίμα να συνεχίζουμε να μιλάμε για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, γιατί το κανονικό θα ήταν να μην χρειάζεται πλέον να συζητούμε αυτό το θέμα. Η μητέρα μου μιλούσε για διαφορές μισθολογικές μεταξύ ανδρών και γυναικών και είναι κρίμα που συνεχίζουμε να μιλάμε σήμερα για το ζήτημα αυτό, αλλά στο σημείο 1 να λέμε ότι δεν έχει γίνει καμία πρόοδος, νομίζω ότι είναι και κάπως υπερβολικό. Θα πρέπει εδώ να ξεβρούμε ένα διαφορετικό όρο, τουλάχιστον στην Ισπανία, όπως έλεγε ε, και η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές ε, υπάρχει ένα σχέδιο για την ισότητα και κάθε έτος βελτιώνεται η κατάσταση των γυναικών και είμαι πεπισμένη ότι σε πολλές χώρες ε, βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Συνεχίζουμε βέβαια να μιλάμε για ανισότητα σε πολλές πτυχές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω βέβαια ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επαναληφθούμε, οπότε δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς θέλω να πω ότι για το σημείο 6 εκεί αναφερόμαστε σε γυναίκες με μεταναστευτικό παρελθόν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, όπως η Ρωμά. Ε, οι Αθήγανες λόγω των οικονομικών τους χαρακτηριστικών έχουν πάρα πολλά προβλήματα για να ενταχθούν στην επαγγελματική ζωή, έχουν δυσκολίες να λάβουν ε, καλύτερη εκπαίδευση και ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να μιλάμε και για αυτές τις γυναίκες σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια όταν αναφέρεται στην ε, ηγετική θέση των γυναικών ε, και επίσης ε, να ενισχύσουμε τη θέση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και τις γυναίκες στο Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν είμαι υπέρ των ποσοστώσεων προσωπικά. Πιστεύω ότι δεν είναι κάτι ορθό ο καλύτερος τρόπος για να κατορθώσουμε να είναι οι γυναίκες να διορίζονται σε υπεύθυνε θέσεις αλλά πιστεύω ότι κατά τα λοιπά είναι πάρα πολύ σωστή η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ. Η κυρία Μωρά, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ναντιαχύρης, ε, αλλά και την κυρία ε, Νεντέλτσεβα για αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική και προσεγγίζει πάρα πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να επιμείνω όμως σε περισμένων σημείων που δεν έχουν τονιστεί επαρκώς και νομίζω ότι πρέπει να τα αναπτύξουμε. Το πρώτο σημείο είναι το πρόβλημα των μισθών. Σήμερα θα πρέπει η Ευρώπη να έχει δεσμευτικούς όρους προκειμένου να ε, υπάρχει ισότητα των μισθών στην πραγματικότητα. Θέλω να μιλήσουμε για πραγματικούς μισθούς, όχι για μείωση του χάσματος, γιατί όλοι σας λένε, κοιτάξτε, ίδιοι είναι μισθοί, το είναι αλήθεια στο δημόσιο και δεν είναι τελικά αλήθεια, γιατί υπάρχει, υπάρχουν αυτά τα πριμ, οι πρημοδοτήσεις που δίνονται και αυτά τα πριμ αυξάνουν το χάσμα. Θέλω να μιλήσουμε δηλαδή για πραγματικούς μισθούς. Ε, η πραγματική ισότητα μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Συνδεδεμένο με το θέμα αυτό είναι το πρόβλημα της φορολόγησης των οικοκυριών. Σε ορισμένες χώρες οι φόροι υπολογίζονται επί των μισθών του κάθε ατόμου. Σε άλλες χώρες ε, φορολογείται το νοικοκυριό και όταν φορολογείται το νοικοκυριό τότε φορολογείται περισσότερο μισθός της γυναίκας. Γιατί σε αυτός έρχεται και να πόκεται πάνω στο μισθό του ανδρός που, μένει, που είναι αποτελεί την αρχική πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό γιατί βρίσκεται ο μισθός της γυναίκας στην ανώτερη κλίμακα τις ε, φορολογίες. Έτσι λοιπόν αυτό αποτελεί αντικίνητρο για τις γυναίκες για να συμμετέχουν στην έργο και κατόπιν ε, θα βρουν ε, μία ή μία απασχόληση κτλ. Έτσι λοιπόν θέλω να παρακαλέσω την κυρία να το έχει αυτό κατά νου γιατί πραγματικά αποτελεί παράγοντα που αυξάνει την απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το δεύτερο σημείο λέγεται στην έκθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε, είναι να καταπολεμήσουμε ε, αυτές τις νοοτροπίες που διαχωρίζουν τα επαγγέλματα σε γυναικεία και ανδρικά. Και εδώ βλέπουμε ότι ε, έχουμε γενιές και γενιές ε, που έχουν αυτή την, ε, όπου τους έχει χαραχτεί αυτή η νοοτροπία. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σημαντικές δράσεις με τους επαγγελματικούς ε, κλάδους. Πρέπει να το χάρη σκεφτείτε τις κατασκευές, όπου ε, στον κλάδο αυτό συνήθως απασχολούνται άντρες. Θα πρέπει να έχουμε προγράμματα και πολιτικές που θα καταπολεμήσουν αυτές τις νοοτροπίες. Βλέπουμε όταν ε, κάποιος πηγαίνει σε διάφορα προγράμματα, Λονάρντο, Κομένιος, Εράσμους, κινούνται τα πράγματα. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να θέσουμε σε εφαρμογή τέτοια προγράμματα για να αλλάξουν νοοτροπίες. Το τρίτο θέμα είναι το θέμα των πτυχίων. Λέγεται ότι ε, προδεύουν οι γυναίκες στην εκπαίδευση και είναι πτυχιούχες, όμως ε, το πραγματικό πρόβλημα είναι τι κάνουν ε, οι γυναίκες με τα πτυχία τους όταν μπαίνουν στην επαγγελματική, στον επαγγελματικό χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ε, δεν ε, ακολουθούν ε, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία την οδό που ακολούθησαν στην κατάρτισή τους και αυτό πρέπει να το δούμε ως επένδυση των οικογενειών. Και αν ε, τελικά δεχτούμε αυτή την κατάσταση, οι γυναίκε δηλαδή να είναι πτυχιούχες, αλλά να μην μεταφράζουν τα πτυχία του στην επαγγελματική ζωή, γιατί δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να συμφιλιώσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, τότε μεγεθύνουμε ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το τέταρτο σημείο. Νάντια, σωστά το λες στην έκθεση. Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, Πρόεδρε. Πρέπει να εισαγαγούμε την ισότητα των εικόνων και στα διοικητικά συμβούλια, αλλά επίσης θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε ε, στο δημόσιο τομέα τα κράτη-μέλη να δώσουν το παράδειγμα. Αν δείτε την πυραμίδα απασχόλησης ε, ανά ε, λειτουργήμα, πάντοτε στα διάφορα κράτη, στην πλειοψηφία των πιο ψηλών θέσεων είναι οι άνδρες και θα πρέπει τα κράτη να δώσουν το παράδειγμα. Ε, δεν αρκεί να επιβάλλουμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να υπάρχει ισότητα, ή αντιπροσώπευση άνδρων και γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια. Θα πρέπει και τα ίδια τα κράτη να το πράξουν αυτό. Σας ευχαριστώ. Τέσσερις ομιλητές έχουν απομείνει. Πάντως ε, πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 9.30. Να είστε σύντομοι σας παρακαλώ. Κύριε Μαν και κατόπιν κυρία Εστρέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν πρέπει να βιαστούμε, να πω τα εξή. Στην ε, Γερμανία ξέρουμε ότι η πρόοδος γίνεται με ρυθμό χελώνας. Ε, αυτό θα διαρκέσει δηλαδή λίγο παραπάνω. Μίλησα με μία γυναίκα πρόεδρο που μας είπε ότι ε, στόχος μας ε, είναι να ε, γίνει περιττή η δουλειά μας, να υπάρχει τόση, τέτοια ισότητα ε, τελικά που να μην έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ε, βλέπουμε όμως ε, για παράδειγμα ότι οι περισσότεροι καθηγητές ε, μαθηματικών, φυσικής λοιπά είναι άντρες, αλλά και οι γυναίκες σημειώνουν μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν συμβολικοί κοινωνικές κινήσεις, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν την ε, κοινωνία, οι οποίες όμως είναι σημαντικές, δηλαδή μια γυναίκα να πάρει μια σημαντική θέση. Ε, το να μιλάμε για την manager της χρονιάς μπορεί να μην είναι ε, να μην είναι μεγάλο βήμα, ε, είναι όμως ε, συμβολικά σημαντικό. Αναφέρθηκε στο ποδόσφαιρο, αλλά είδα έναν τίτλο ότι ο αθλητισμός γίνεται γένους θηλυκού. Έχουμε δει την ποδοσφαιρίστρια της χρονιάς προέρχεται από τη δική μου πόλη και και ε, σίγουρα ε, ε, εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω το πρωτάθλημα γυναικείου ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Στρέλα και μετά η κυρία Φιγκερέρο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι αναφέρεται στα ουσιαστικά σημεία η έκθεση φυσικά. Ορισμένα σημεία χρήζουν βελτίωση. Η κατάσταση των ε, γυναικών ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια δεν ε, είναι ισότιμη ποικίλη ένα κράτος μέλος και αναφέρομαι και στο ποσοστό συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, και σε ό,τι αφορά τη μισθολογική διαφορά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, κράτη-μέλη όπου η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών φτάνει και στο 30%. Αν και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 18% και επίσης υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την πρόσβαση ε, σε θέσεις πιο σε λήψεις αποφάσεων είτε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό πλαίσιο. Και γι' αυτό θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σημασία της ποσόστοσης. Γιατί παρόλο που η ποσόστοση είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να είναι προσωρινό, ένα εργαλείο που αρνούνται ορισμένε γυναίκες γιατί θεωρούν ότι δεν τους προσδίδει κύρος. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το μέσο αυτό έχει αποκαλυφθεί ως το μόνο που έχει αποφέρει αποτελέσματα. Οι χώρες που ήδη έχουν υιοθετήσει νόμους ισότητας στην πολιτική εκπροσώπηση έχουν έχουν ε, ισορροπία ε, με την εκπροσώπηση των γυναικών ε, είτε στα εθνικά κοινοβούλια είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να υιοθετηθούν ποσοστώσεις για τα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων και για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Νορβηγίας. Και θέλω να επενθυμίσω ότι μια συντηρητική κυβέρνηση στην Νορβηγία ήταν αυτή η οποία έθεσε την ποσόστοση 40% για την εκπροσώπηση των γυναικών στις δημόσιες επιχειρήσεις και για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όχι για οδεολογικούς λόγους αλλά για λόγους οικονομικών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία στην Νορβηγία επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις ε, όπου στα διοικητικά του συμβούλια τουλάχιστον συμμετέχουν τρεις γυναίκες έχουν καλύτερα αποτελέσματα και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Μιλάμε μάλιστα και για αύξηση της τάξης του 72%. Για να μην μακρηγορήσω, θέλω να αναφέρω και μία ακόμη πτυχή που έχει να κάνει με τη συμμετοχή των γυναικών με μικρά παιδιά στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες με παιδιά κάτω των 6 ετών έχουν περισσότερες δυσκολίες να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους και συμμετέχουν λιγότερο στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, οι όμοι με μικρά παιδιά έως 6 ετών σημειώνουν ε, πιο εύκολη πρόοδο, πιο εύκολα πρόοδο και μπορούν ε, να εργάζονται και για περισσότερες ώρες. Έτσι λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικό να υιοθετηθούν μέτρα που να προωθούν τη συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματική ζωής, προκειμένου και οι άνδρες και οι γυναίκες να μπορούν να αναλάβουν Ευθύνε και σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό. Λυπάμαι μόνο που... Και τελειώνω, Πρόεδρε. Λυπάμαι μόνο που στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 όλα αυτά τα σημεία έχουν παραλυφθεί. Τίποτα δεν αναφέρεται σχετικά με την αναγκαιότητα καταπολέμησης της ε, διαφοράς, της μισθολογικής διαφοράς και για την πρόθεση πολιτικών συμφιλίωσης μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση που φυσικά δεν μπορεί να είναι πιο μικροσκελής λόγω του κανόνα για το όριο των λέξεων και των χαρακτήρων, μπορεί να συμπληρωθεί Τώρα με κάποια θέματα που εγώ θεωρώ σημαντικά. Και εγώ θα συνεισφέρω μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε τις πολιτικές ε, λιτότητας ε, οι οποίες επιδεινώνουν τις διακρίσεις και είναι πάρα πολύ αρνητικές για τις γυναίκες ιδίως και για τα παιδιά γιατί επιδεινώνουν ε, την ε, επισφαλή εργασία και την κακοπληρωμένη εργασία, την ανεργία και επίσης αυξάνονται και οι μισθολογικές διαφορές. Ε, ακόμη έχουν επίπτωση στη φτώχεια, στις κοινωνικές παροχές που παρέχονται. Έχουν λοιπόν πολύ ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών και ε, σημαίνει ότι έχουμε επαναχώρηση στην εφαρμογή των δικαιωμάτων. Κάτι ακόμη θέλω να πω ότι η μισθολογική διάκριση σημαίνει ότι υπάρχει και διάκριση στις συντάξεις και σημαίνει ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες στα γυρατιά και χειρότερες συνθήκες ζωής για τις ηλικιωμένες γυναίκες και φυσικά και σε αυτό πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή αυτή τη στιγμή που η φτώχεια των γυναικών αυξάνεται. Και ε, φυσικά αντικατοπτρίζεται κατόπιν και στα παιδιά. Και σε μια Ευρώπη που είναι όλο ένα και λιγότερο κοινωνική. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Κονέλησεν, θα ήθελα να τονίσω την θετική πλευρά, της πολλές τροποποιήσεις που γίνονται, τις πολλές αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ε, μπορούμε να αδράξουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τις ε, πολιτικές προς όφελος των γυναικών. μια αλλαγή προς μια πιο πράσινη οικονομία. Ε, είναι μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε οι γυναίκες να μην μείνουν πίσω στην μεταβατική αυτή περίοδο. Και η στρατηγική Ευρώπη 2020 σημαίνει ότι πολύ περισσότερος κόσμος στην αγορά εργασίας ε, μπορεί να ε, ότι πολύ περισσότερο κόσμο μπορεί να δουλέψει στην αγορά εργασία, γιατί το μεγαλύτερο δυναμικό στην αγορά εργασία αυτή τη στιγμή, που, το οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε, είναι οι γυναίκε. Θα μπορούσαμε να του δώσουμε, για παράδειγμα, δικαίωμα στην ε, ε, μερική απασχόληση ε, και να κάνουμε ρυθμίσεις για να υπάρχει φροντίδα των παιδιών. Το να τα αφήσουμε όλα στους κοινωνικούς εταίρους ε, είναι κάπως ανησυχητικό, διότι έτσι ε, μένουμε εκτός εμείς. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Όσον αφορά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, αυτό είναι κάτι που γίνεται σε μεγάλη κλίμακα αυτή τη στιγμή λόγω της οικονομικής κρίσης. Ε, θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία αυτή για να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών στις ε, θέσεις ηγεσία. Συμφωνώ με την κυρία Εστρέλα ότι είναι απαραίτητες οι ποσοστώσεις, ε, αν και ως προσωρινό μέτρο. Γνωρίζουμε ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι καλό πράγμα για τις γυναίκες, διότι θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τα προσόντα τους. Τίποτα άλλο όμως δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Εάν τα τελευταία 30 χρόνια ο αριθμός των γυναικών στις σχετικές θέσεις δεν αυξήθηκε, γιατί να αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια ε, ε, εάν δεν λάβουμε μέτρα όπως είναι οι ποσοστώσεις. Ποτέ ε, δεν άκουσα άντρα να παραπονιέται ότι ε, τον επιλέξανε για μια θέση καλή επειδή είναι άντρα, ε, ενώ αυτό γίνεται πολύ συχνά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Άτια Χίρσου να απαντήσει, αλλά ε, λίγο σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ναι θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που έγινε, για τις πολύ καλές προτάσεις που ακούσαμε. Όπως ε, ήδη είπα, θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες. Ε, περιμένω να δω και τις τροπολογίες των σκιωδών εισηγητών, καθώς και των άλλων μελών. Ε, εγώ εδώ έχω αναφέρει κάποια πράγματα, αλλά μπορεί οι συνάδελφοι να με βοηθήσουν ε, να ε, βελτιώσουμε τα σημεία αυτά. Ίσως πίνοντας ένα καφέ μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σύντομοι. 9 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία της τροπολογίας, 24 Ιανουαρίου η συζήτησή τους και 25 Ιανουαρίου η έγκριση. Ε, προχωράμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι θα ψηφίσουμε μαζί. Unblock υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία μας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 κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις 23 υπέρ, 17 κατά δείχνει εδώ, αλλά και κάποιος που έχει ξεχάσει κάρτα, τώρα 18, 22 καταπίπτει, 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ, κατά, αποχές,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 εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 52 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 24 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβιβαστική σίγματα F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G ζήτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Καταπίπτουν αφού εγκρίθηκε η συμβαστική. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 αποσύρεται. 78. Α, μια στιγμή θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Όσον αφορά την τροπολογία 78, θέλουμε μια διευκρίνηση, διότι υπάρχουν διαφορές ε, στις ε, στην ε, αγγλική και γερμανική εκδοχή. Θέλουμε στα αγγλικά το piracy να το αντικαταστήσουμε με το counterfeiting. Αν δεν έχει κανείς αντίρρηση, όχι, καλώς. Με την αλλαγή αυτή, 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για την 81. Ξεκινάει η ψηφοφορία λοιπόν. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ακόμα. Α, μπορούμε να ψηφίσουμε. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες. «22 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται». 71 κατά 80 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε και για την 80. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες. «23 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση, αλλά με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 38 υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Στην εισηγήτρια. Η επόμενη ψηφοφορία τώρα είναι το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Παπαδοπούλου. Η κυρία Φιγκερέδο θα πει κάτι όταν φτάσουμε στη συμβιβαστική Δέλτα. Συμφωνεί. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση της κυρίας Παπαδοπούλου που είναι σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων ε, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-2013. Ε, τροπολογία 1, υπέρ. Α, ζητήσατε αν μπλοκ να ψηφίσουμε την 1 μέχρι και 9. Συμφωνείτε? Υπάρχουν προβλήματα. Α, 1 με 8. Εντάξει. Συμφωνεί. Ωραία, αν μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά Αποχές. Νομίζω το απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 20. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. 24 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για την 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Τροπολογία 29. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. 25 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και πάλι. 31. Τροπολογία 31. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 24 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε. 32 λοιπόν, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 24 υπέρ 16 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Δέλτα. Δι. Κυρία Φίγερε εδώ. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Σε αυτό το συμβιβασμό είχε συμπεριληφθεί η δική μου τροπολογία 37. Εγώ συμφωνώ να βρίσκεται εδώ, όμως η προηγούμενη εκδοχή ε, είναι αυτή η οποία πρέπει να ψηφιστεί. Εγώ όμως έχω αντιρρήσει σε σχέση με το πρώτο τμήμα του συμβιβασμού, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ψηφοφορία μας. Έτσι λοιπόν εμείς θα έπρεπε να ψηφίσουμε την πρώτη εκδοχή του συμβιβασμού και όχι αυτή που μας στάλει σήμερα που αποσύρει την τροπολογία μου αλλά δεν τη συμπεριλαμβάνει ως ξεχωριστή ως ξεχωριστό τμήμα προς ψήφιση. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να προτείνω στην εισηγήτρια να ψηφίσουμε τη συμβιβαστική πρόταση που είχαμε χθες και όχι αυτή που εστάλει σήμερα. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική ω έχει. Τώρα αν λέτε ότι δεν καλύπτεται καθόλου η δικιά σα τροπολογία από το συμβιβασμό, τότε θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την τροπολογία σα 37 επιπλέον ως προσθήκη στο συμβιβασμό. Εφόσον συμφωνούν όλοι. Έτσι, ωραία. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 37 ως προσθήκη Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη, Ωραία. 40 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ή υπέρ, κατά, να ελέγξουμε για τη συμβαστική ε παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. 26 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Δύσκολο αυτό. Ας ελέγξουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. 48. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Εγκρίνεται. Συμβαστική F ταφ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ελέγχουμε για την 56. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της προφορίας. 24 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε πάλι παρακαλώ. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 57. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. 22-21 είναι το αποτέλεσμα. 22 υπέρ, 21... Α, όχι, ανάποδα, ανάποδα λέει η πρόεδρος. 21 ψήφι υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την ε, τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Σαράντα υπέρ, δύο κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. προχωράμε στην τελική ψηφοφορία που έχουμε. Σχέδιο έκθεσης για την ε, του Λούντιξεν ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Δεν νομίζω ότι σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, ε συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 7 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία, την τροπολογία 7, αρχή της ψηφοφορίας. Everyone Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική τροπολογία Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 12, αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C, γ, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Χωριστή ψηφοφορία έχει ζητηθεί για την τροπολογία 18. Πρώτο μέρο υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το πρώτο μέρος της τροπολογίας 18, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές το ίδιο εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά Πολύ μικρή η διαφορά, να ελέγξουμε. Ε, αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 20. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Το ίδιο. Απορρίπτεται. 22. Είναι συμβατή με την 21. Ε, τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 22. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 υπέρ. Συγγνώμη, 20 υπέρ. 22 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. μαζί με την 24. Ε, διαγραφή υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε για να είμαστε βέβαιοι. Ελέγχουμε λοιπόν για την τροπολογία 23 και 24. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 11 υπέρ, 30 κατά. Δεν ήταν και τόσο μικρή διαφορά. Ε, ε, συμβαστική δέλτα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 έχει αποσυρθεί, 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έτσι τελειώνουν οι ψηφοφορίες μας. Να προχωρήσουμε στη συζήτηση σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και τι πολιτικέ συνέργειες για την αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακής Αναπτυξη και άλλων διασφαλιστικών ταμείων. Να δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπω γνωρίζουν στα αδελφή κοινωνική συνοχή, όπω και δευκή συνοχή, είναι όχι μόνο θεμελιώδη αρχές τη πολιτικής της Ένωση, αλλά και ε, τους πλέον ε, και σημαντικούς παράγοντες. Συγγνώμη, παρακαλώ, όσοι αποχωρείτε, σας παρακαλώ, όσο πιο σιγά μπορείτε, γιατί ο κ. Κονφεράτη έχει δει πάρει το λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι η διαφυγή συνοχή και ε, η πολιτική συνοχή είναι θεμελιώδεις πολιτικές της Ένωσης, αλλά αποτελούν και παραγόντες ανταγωνιστικότητας, ε, όπως φάνηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επικράτες είναι σε θέση να προσελκύσουν ε, επενδύσεις όταν συνοδεύονται από στοιχεία συνοχής και κατόπιν έχουμε διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας που είναι απαραίτητες για να έχουμε ποιοτικά προϊόντα που να ανταγωνίζονται παγκοσμίω. Πρέπει λοιπόν ε, να ολοκληρωθεί η συνοχή και αυτή η ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι παρά να είναι μια αξιόλογη ανάπτυξη με ισομερή μέτρα ε, στην επικράτεια και που θα διασφαλίζουν την ευημερία των ατόμων βάσει και τις δημιουργίες νέων θέσεων εργασίας αυτά τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης είδαμε πως τα διαφορετικά ταμεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δυστυχώς ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο. Δυστυχώς ένα τμήμα των διαθέσιμων πόρων ε, χάθηκαν, διασκορπίστηκαν, ενώ άλλοι πόροι δεν χρησιμοποιήθηκαν ε, καταλήλως και δεν χορηγήθηκαν σε όποιον του ζήτησε. για την υλοποίηση στρατηγικών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο που αναφέρονται στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 πολιτική κοινωνική συνοχή είναι αυτή, και αυτή της εδευτικής συνοχής πρέπει να συντονιστούν και να συνδεθούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Γιατί βλέποντας ε, τι έγινε στο παρελθόν, μπορούμε να δούμε ότι δεν υπήρχε πάντοτε συντονισμός και η έλλειψη συντονισμού και στην ίδια την επικράτεια οδήγησε σε μειωμένη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ε, των ταμείων της Ένωσης, των κονδυλίων από την Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε την κοινωνική συνοχή με τις δράσεις που ε, προκύπτουν από την εδαφική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο όμως πρέπει με προσοχή να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στις δραστηριότητες που οδηγούν σε μια ποιοτική απασχόληση, αναφέρομαι στη στην κατάρτιση, στις διαδικασίες έρευνας και κοινοτομίας. Αλλά το κοινωνικό ταμείο σε αντίθεση με μια διαδεδομένη άποψη, ακόμη και στο κοινοβουλίο μας, κατά την άποψή μας θα έπρεπε να διατηρηθεί ως ε, βοηθητικό μέσο. Ένα είναι να καθορίζουμε το συντονισμό, να μιλάμε για συντονισμό μεταξύ των ταμείων ε, και διαφορετικό είναι να καταργήσουμε εντελώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όπως ζητούν ορισμένοι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει ως στόχο να ε, καθιστά καλύτερη την ποιότητα της εργασίας, αλλά αυξάνει και την ποσότητα των θέσεων εργασίας. Πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν. Πρέπει να φτάσουμε λοιπόν σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα Πρέπει να διαχωρούμε το ΕΚΤ από τα υπόλοιπα κίνητρα. Ακόμη και τα μέτρα ε, απόκλησης χρειάζονται αυτή τη διάκριση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εισαγάγουμε κανόνες που θα επιτρέπουν ε, στις ε, περιφέρειες να έχουν καλύτερο έλεγχο και από τη δική μας σκοπιά να επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν να εμπλέξουν όχι μόνο τις περιφέρειες αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλους τους stakeholders οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη χρήση του ΕΚΤ. Έτσι λοιπόν, Πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να παρουσιάσει γρήγορα μια μεταρρύθμιση των διαφορετικών ταμείων, έχοντας ε, όμως ε, διατηρώντας ε, και κατά νου όλα τα θέματα που αφορούν την απασχόληση και πρέπει η απασχόληση να είναι κεντρικό σημείο στη στρατηγική το 2020. Επί της ουσίας, ε, αυτό είναι το νόημα της δικής μου πρότασης. Δηλαδή, σημειώνουμε τις δυσκολίες ε, που εντοπίσαμε στη χρήση των ταμείων. Να λάβουμε υπόψη την τεράστια αξία που έχουν τα ταμεία ως συνιστώσεις για τη στρατηγική 2020, να ζητήσουμε αναδιοργάνωση, αλλά στο εσωτερικό αυτής της αναδιάρθρωσης να διατηρήσουμε τη διάκριση σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσπαθώντας ε, να ε, ε, εμπλέξουμε και τις περιφέρειες και τους stakeholders. Φυσικά θέλω να δω ποια είναι η άποψη και των συναδέλφων και φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμη πιο ρητές οι παρεμβάσεις του και μέσω της τροπολογίας και φυσικά θα τις εξετάσω και θα επανέλθω και θα ξανασυζητήσουμε μαζί όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ανέφερε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι ε, μια συνταγή επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολύ συχνά κάνουμε ένα σωρό μελέτε, ε, τελικά όμω δεν φτάνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει. Ενώ με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, μπορούμε έτσι να ε, αντιμετωπίσουμε την κρίση, στηρίζεται η απασχόληση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ε, είναι ε, ένα στοιχείο ποιότητας. Μιλάμε για ποιότητα και για ποσότητα στην έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη αναφέρει ότι θέλει ενιαία ε, διαχείριση. Ε, θέλουμε συντονισμένη, όχι όμως ε, απόλυτα ενιαία. Θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν υπάρχει συντονισμός στις διάφορες χώρες, αλλά όχι να καλύπτει μια μεθοδολογία όλα. Συμμερίζομαι δηλαδή απόλυτα τη βασική ιδέα. Πολλοί είπαν ότι πρέπει να ε, απλοποιηθούν τα πράγματα ε, και όλα αυτά να υπόκεινται στην Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτό θα πρέπει να το εμποδίσουμε. Σίγουρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί η βασική ιδέα και γι' αυτό πράγματι συμφωνώ έτσι με τις περισσότερες ιδέες σου. Ε, μπορεί να θέλω να υποβάλω δύο-τρεις ε, τροπολογίες, ε, πιο πολλοί όμως έχουν χαρακτήρα επιβεβαίωσης αυτών που λες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την έκθεσή του. Η αποφασιστική παράγραφος είναι η παριθμόν 7 και νομίζω ότι ε, αυτή ακολουθεί αυτό που έχουμε αποφασίσει. Ε, θέλουμε τα ταμεία να καλύπτονται από έναν κανονισμό αλλά να έχουν ξεχωριστούς κανόνες. Δυστυχώς στην ε, ψηφοφορία απορρίφθηκε μια σημαντική τροπολογία δική μου. Είναι η τροπολογία που αναφέρει τις εξελίξεις ε, των τελευταίων ε, μηνών. Έχω την εντύπωση ότι δεν πέρασε επειδή δεν ήταν πολύ σαφής η μετάφραση επειδή δεν το συζητήσαμε αλλά θέλω να πω ότι εάν ε, συνεχίσουμε με τον ε, τρόπο που προχωράμε τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα λαμβάνει όλο και λιγότερα χρήματα. εδώ σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο ε, καθορίζουμε εμεί ε, τι ποσοστό των διαφορετικών ταμείων θα πρέπει να εισρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, αυτό θα πρέπει μήπως να το αφήσουμε στα κρατημέλη. Αυτή είναι πολύ δύσκολο ερώτημα και είναι ασαφές αυτή τη στιγμή. Πάντως θα πρέπει σίγουρα να το συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, το επόμενο ερώτημα είναι ότι ε, η Επιτροπή των ε, Περιφερειών ε, και η αρμόδια Επιτροπή. αυτό μας ενδιαφέρει πολύ το πώς αποφασίζονται τα πράγματα εκεί. Ε, είμαι ευγνώμων που η, ε, που ο συγητή λέει σε μια από τι πρώτε παραγράφου ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, πολιτική συνοχή. Χρειαζόμαστε ε, και τον κοινό κανονισμό, ο οποίο να καλύπτει και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιτροπή. Γι' αυτό ε, ήδη κατά τον ε, κανονισμό με ενδιέφερε ε, να καλύπτει ο κανονισμός όλα τα ταμεία, αλλά να μην υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στα ταμεία. Το επόμενο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην συζήτηση για την πολιτική συνοχής. Ε, και οι κανόνες για τον έλεγχο. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να μην είναι εις βάρος των προγραμμάτων. Ε, ο, μεγάλος, ε, ο γενικός κανονισμός θα καλύπτει όλα τα ταμεία, θα έχει να κάνει και με το ΦΠΑ, θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να βρούμε μια καλή διατύπωση. Θα το θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτό περαιτέρω. Πάντως αυτά είναι τα βασικά ε, τρία ζητήματα τα οποία αν δεν περάσουν θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Λίζα Μπεθέρς. Απροηγουμένως κύριε Ευχαριστώ. Η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και κυρίως, και κυρίως τον κύριο Τόμας Μαν για αυτά που είπανε για την έκθεση του συναδέλφου Κομφεράτη. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πολιτικές συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι πραγματικά ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να θέσουμε τους κανόνες και τους άξονες. Πρέπει να είναι ορατές οι πολιτικές αυτές και πρέπει η κοινοτική αυτή προσέγγιση να αποτελεί τον κανόνα και έναν κανόνα εύκολα κατανοητό και ορατό. Δεύτερον, σημείο 7. Στο σημείο 7 αναφέρεται. Σύμφωνο απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι είναι αναγκαίο να διακρίνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από αυτά. Να είναι πολύ συγκεκριμένο το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό το οποίο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά τους κατοίκους ε, περιφερειών που έχουν ανάγκη από το Ταμείο Συνοχής. Τρίτο σημείο. Πρόκειται για την παράγραφο 8. Όταν συνεδριάζουμε επιτόπου και συναντιόμαστε με την αυτοδίκηση, μας ε, ζητούν συνέχεια πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή τους και διαπιστώνουμε ότι δεν γνωρίζουν πολλά για την χρηματοδότηση που μπορούμε να προσφέρουμε και το άλλο που μας λένε είναι ότι πάντα δυσκολεύονται με τη γραφειοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να απλοποιήσουμε. Ναι, μεν έχουμε αυτή την ε, ευρεία διάσταση, αλλά από την άλλη μεριά να φροντίσουμε να είναι εύκολη η χρήση των κονδυλίων. Απλούστευση λοιπόν της διαδικασίας. Εγώ επιμένω γι' αυτό. Όταν πηγαίνουμε επί τόπου, ειλικρινά αυτό μας ζητάει η αυτοδίκηση. χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αντίφαση με το τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας. Και αυτό είναι το εξή. Συχνά είναι οι ίδιες οι περιφέρειες οι οποίες εποφελούνται από το Ταμείο Συνοχής και που οι ίδιες προσθέτουν γραφειοκρατία ή βάζουν άλλου πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι τελικά τροποποιούν, αλλάζουν την κοινοτική πολιτική. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Δηλαδή, μια υπερβολή αποκέντρωσης των κονδυλίων αυτών και του ΦΕΝΤΕΡ και του Κοινωνικού Ταμείου εμποδίζουν την προβολή της Ευρώπης επιτόπου και τροποποιεί την ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική που θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε όσον αφορά τη συνοχή. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, όχι απέναντι στους χρήστες, αλλά πιο αυστηροί απέναντι στους ενδιάμεσους, που είναι οι περιφέρειες και οι οποίες περιπλέκουν την διευκόλυνση αυτή που προσφέρουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα κύριε Χέρση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολλά σημεία ήδη αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Μαν και την κυρία Σρέτερ. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το μέσο μας για να ασκούμε πολιτική απασχόλησης ε, και αγοράς εργασίας. Είναι ακριβώς το μέσο το οποίο βλέπουν οι πολίτες όταν υπάρχει μια ταμπέλα που λέει ε, προωθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σημαντικό είναι η ε, σχετική αρμοδιότητα να παραμείνει στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Εννοείται ότι θα υπάρχει συντονισμός με άλλα ταμεία όπως είναι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι λογικό. Κατά τα άλλα θα είχαμε τελείως ανεύθυνη πολιτική αλλά είναι δικό μας μέσο και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να ασκούμε με αυτό πολιτική. Θα πρέπει όμως επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι σε κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ε, ομάδες ε, μειονεκτικές και οι οποίες μπορούν να υποφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και σε πλούσια κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη οι μικρές τοπικές ενώσεις εξαρτώνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να ε, βοηθούν κάποιες ε, ομάδες πληθυσμού τους, ε, νέους, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες κλπ. Θα ήθελα Λοιπόν, να συνεχίσει να είναι δυνατή η απόδοση πόρων σε όλα τα κράτη-μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν έτσι να δείξουμε προ ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε εμεί η Επιτροπή απασχόληση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι θα πρέπει να ε, διατηρηθεί η αρμοδιότητα του Ταμείου στην Επιτροπή απασχόληση. Ε, και ξέρω ότι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θέλει να το αναλάβει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μα, ώστε να φροντίσουμε να παραμείνει εδώ η αρμοδιότητα. Ο κύριο Κοφεράτη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Είμαι πολύ καροποιημένος που το θέμα της διάκρισης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τα υπόλοιπα θεωρείται κεντρικό ζήτημα από όλους. Δεν ε, είχα αμφιβολίες ότι αυτή ήταν ε, η άποψη που υπερίσχε στη δική μας Επιτροπή. Γιατί η αντίθετη άποψη που όπως γνωρίζετε είναι βαθιά ριζωμένη και στο Κοινοβούλιο, θα μπορούσε ε, ε, να αναχαιτιστεί αν εμείς συμφωνήσουμε επί του σημείου αυτού. Φυσικά και θα εμπλουτιστεί το κείμενο, αλλά το κεντρικό ζήτημα είναι αυτό και επί αυτού πρέπει να συγκλίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοιου είδου ευαισθησία στην Επιτροπή για προφανούς λόγους. Δεν βλέπω διαφοροποίησεις ε, μεταξύ πολιτικών ομάδων. Πρόκειται για διακρίσεις που γίνονται από το λειτουργήμα του καθένα. Όσοι διαχειρίζονται τις ε, τις ε, δαφικές πολιτικές έχουν την τάση να τα βάζουν όλα μαζί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα. Εμείς ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά και η ποιότητα της δουλειάς. Και αυτό το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου. Οι περιφέρειες και οι ε, περιφερειές πολλές φορές τείνουν ε, να ενοποιούν τις πηγές, να τις ομογενοποιούν και κατόπιν αυτοί αποφασίζουν τι πράττουν ε, ε, ανάλογα και με την προέλευση της χρηματοδότησης και το κάνω και γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλος έλεγχος. Ε, αυτή η πολιτική μάχη πρέπει να δοθεί από εμά, γιατί αν το ΕΚΤ γινόταν ε, ένα μέσο αδιαφοροποιητό, εγώ νομίζω ότι η στρατηγική για το 2020 θα δικαιβευόταν. Είναι ένα καθόλου απλό ζήτημα, γιατί Βλέπουμε εδώ πολλούς συναδέλφους να προωθούν μια μεταρρύθμιση που ε, ακυρώνει την αυτονομία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας δούμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες 14 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. 24-25 ε, θα έχουμε συζήτηση και πριν του Φεβρουαρίου θα έχουμε την υιοθέτηση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τώρα και αυτό το σημείο. Θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση για, τα... για το μηχανισμό μικροχρηματοδότησης. Θα κάνουμε διάλειμμα 5 λεπτών έτσι ώστε να μπορούν να έλθουν και οι εμπειρογνώμονες. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλο το πάνελ θα βρίσκεται εδώ και θα αρχίσουμε και πάλι στις 10.30. Θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά. Ετοιμαστείτε. Uh, thank you. And I Καλωσορίζω τους ε, εμπειρογνώμονές μας εδώ. Έχουμε τέσσερις προς το παρόν και περιμένουμε ακόμα έναν που θα έρθει. Όπου να είναι φαντάζομαι ο καιρός θα φταίει. Όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα στις χώρες μας. Θα ζητήσω όμως πρώτα απ' όλα την κυρία Μπρουλιόνο να μιλήσει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Αλλά όχι, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος. Προηγουμένως η Κίνγκα Γκόντς. Παρακαλώ, η Κίνγκα Γκόντς θα πάρει πρώτα το λόγο και μετά θα περάσω στους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη εισαγωγή, η οποία θα περιέχει περισσότερο ερωτήσεις για τις οποίες θα θέλαμε να ακούσουμε απαντήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να έχουμε αυτήν την ε, δημόσια ακρόαση τόσο νωρίς μετά την λήψη της σχετικής απόφασης για να δούμε πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Θα ήθελα να φέρω κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού που θεωρούμε πολύ σημαντικά. Πιστεύουμε ότι είναι ε, σημαντικό, ε, διότι όταν το ετοιμάζαμε υπήρχε μια αίσθηση του επιγόντος ε, Θεωρήσαμε ότι είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ευέλικτο και ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πρώτων συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την πτυχή της εφαρμογής είχαμε μια βιντεοδιάσκεψη και είχα την εντύπωση ότι υπάρχει Υπάρχουν καθυστερήσεις ε, και βρισκόμαστε ακόμα στην προκαταρτική φάση. Βρισκόμαστε ήδη στο 2011, ενώ εμείς ελπίζαμε να ξεκινήσει η πραγματική λειτουργία, η ουσιαστική λειτουργία του προγράμματος το 2010 ήδη. Η Κομισιόν ε, υποσχέθηκε και ήταν και ελπίδα μας η φύση αυτού του ταμείου να προσελκύσει περισσότερους πόρους. Η εκτίμηση ήταν να έχουμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, μέρος των οποίων θα προερχόταν από εμπορικές τράπεζες. Από ό,τι ξέρω από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, είναι πολύ μικρότερο το ποσό που έχουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά με το πώς ε, σκοπεύετε να συγκεντρώσετε περισσότερους πόρους από ε, εμπορικές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει κυρίως τον κίνδυνο και αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις εμπορικές τράπεζες. Είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση, είχα προγραμματίσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία όμως βλέπω ότι διαγράφει τελικά από το πρόγραμμα. με βάση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήταν ενδιαφέρον να εντοπίσουμε ποιοι χρειάζονται περισσότερο την ε, οικονομική αυτή βοήθεια. Ε, αναζητήσαμε την, επιδιώξαμε να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία και θέλαμε να ξεκινήσουμε από δύο χώρες ε, που έχουν καλό ιστορικό. Το Επενδυτικό Ταμείο και η Κομισιόν, από ό,τι ξέρω, ετοιμάζει συμβάσεις ε, με άλλες χώρες επίσης. Ε, και μάλιστα χώρες που έχουν και αυτές τέτοιο ιστορικό και που είναι έτοιμες να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα προχωρήσετε και πέρα από αυτό όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία δηλαδή. Το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε το στοιχείο της καθοδήγησης, το οποίο δεν καλύπτεται από το Ταμείο. Και από ό,τι βλέπω, δεν ε, υπάρχει ακόμα κάποια εγγύηση για κάλυψη του στοιχείου αυτού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω πώς ε, σκοπεύετε να διασφαλίσετε το στοιχείο αυτό, το οποίο είναι το πιο βασικό ε, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα από τους ε, συνήθεις ε, πελάτες της ε, οικονομικής βοήθειας. Να προχωρήσουμε στους ανέργους, για παράδειγμα, που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Πολλοί από τους πιθανούς πελάτες δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω και εδώ πώς ε, σκοπεύετε να προχωρήσετε και να διαδώσετε τις πληροφορίες. Ε, και το βασικό ερώτημα, νομίζω για όλους μας με βάση τις προηγούμενες ε, συζητήσεις, είναι πώς μπορεί αυτό το νέο μέσο να επικεντρωθεί στις ε, μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες και χώρες και να μην εφαρμόζεται στα ε, ήδη ε, ε, καλά ανεπτυγμένα συστήματα μικροχρηματοδότησης. Πώς δηλαδή θα αποφύγουμε να έχουμε απλά άλλο ένα μέσο το οποίο να στηρίζει μια οικονομικά βιώσιμη μικροαστική τάξη. Ελπίζω να ακούσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλους όσους συμμετέχουν από την πλευρά του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα περάσουμε στον πρώτο πυρογνώμον από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Λουξεμβούργο. Είναι η κυρία Μπρουν Λεόν. Για 10 λεπτά παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ σήμερα και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την δημιουργία του Progress Microfinance Instrument. Εγώ εκπροσωπώ το μέσο αυτό και θα ήθελα να σας βοηθήσω να καταλάβετε τις ε, βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τα καλά αποτελέσματα που έχουμε ήδη πετύχει. Πιστεύω ότι θα δώσω απαντήσεις στις ερωτήσεις της κυρίας Γόντς. Πρώτα απ' όλα, μπορώ να σας πω ότι το δεύτερο τμήμα της πιστοτικής διευκόλυνσης έχει ήδη ξεκινήσει και ότι πολύ συγκεκριμένες δράσεις βρίσκονται στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να θυμηθούμε το πολιτικό πλαίσιο μοναδικό αυτή τη στιγμή μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις αλλά και για τους ε, ανεξάρτητους εργαζομένους έτσι ώστε να βοηθήσουμε ε, άνεργους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας ή να μπουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά. Προσπαθούμε να τους συμπεριλάβουμε τελικά στο συμβατικό τραπεζικό τομέα. Οι επιπτώσεις της πρωτοβουλίας αυτές ε, πρέπει να είναι ορατές πολύ γρήγορα αλλά πρέπει να έχουν και μεγάλο εύρος. Με πέντε φορές το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε η Κομισιόν, που φτάνουν σε μικροδανιστές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον όμως, από τον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, η διευκόλυνση αυτή, η πιστοτική αυτή διευκόλυνση, αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο και για την παρετέρω πρόθεση της αγοράς μικροπιστώσεων προκειμένου αυτή να είναι βιώσιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια συγχρόνως, ότι από μόνη τη η πιστοτική αυτή διευκόλυνση, οι μικροπιστώσεις δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Ούτε είναι δυνατόν η Progress Microfinance ε, να ε, αποτελέσει τον μόνο καταλήτη που θα βοηθήσει σε παρετέρω ανάπτυξη της ε, ευρωπαϊκής αγοράς μικροπιστώσεων. Επιπλέον χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να βοηθήσει να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα μικροπιστώσεων. Είναι και αυτά δηλαδή εξίσου σημαντικά. Για παράδειγμα, πώς θα καλύπτεται το κόστος των ε, ενδιάμεσων χρηματοδοτικών ε, φορέων και πώς θα έχουμε πόρους για την οικοδόμηση ικανοτήτων. Είναι μερικά παραδείγματα αυτά. Οι υπεύθυνοι που δημιούργησαν την διευκόλυνση αυτή αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις ήδη από την αρχή. Ε, ξεκινώντας ε, θα σας πω τη δουλειά που έγινε όσον αφορά την ε, ανάπτυξη που έπρεπε να βοηθήσει και τους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς. Αναπτύξαμε λοιπόν μια στρατηγική έτσι ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε και την κοινωνική διάσταση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τότε σε ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή βάση. Επιπλέον, από τη στιγμή που η αγορά η ευρωπαϊκή μικροπιστώσεων είναι πολύ διαφοροποιημένη, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία λύση για όλα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα και μόνο προϊόν που θα μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Αντίθετα, χρειαστήκαμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων για να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες των διάμεσων χρηματοδοτικών φορέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος, όντως, γιατί έχουμε ε, περιπτώσεις που έχουν πολύ έντονη την κοινωνική διάσταση, όπως είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως έχουμε και εμπορικά προσανατολισμένα όργανα, όπως είναι οι εμπορικές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα θα σας δώσω ένα παράδειγμα ένα μικροπιστωτικό ίδρυμα στην Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο μια στήριξη μακροπρόθεσμα, μια χρηματοδότηση μακροπρόθεσμα. Αν όμως δείτε μια άλλη startup ε, κοινοπραξία ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Δυτική Ευρώπη, αυτή αντίθετα χρειάζεται ένα δυνατό αρχικό κεφάλαιο. Οι εμπορικέ τράπεζε από την άλλη μεριά δεν θέλουν πολλού περιορισμού για να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε καλή τιμή αλλά μπορούν να υποφεληθούν περισσότερο από μια εγγύηση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση στις ανάγκες, γι' αυτό και εμείς φροντίσαμε να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών μέσων μικροχρηματοδότησης, είτε είναι δάνεια, είτε είναι συμμετοχή στο κεφάλαιο, είτε είναι εγγύησης. Και αυτό είναι πολύ βασικό για να πετύχουμε ε, κάτι καλό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, το μεγάλο εύρος αυτό προϊόντων απαιτεί και διαφορετικά σχέδια εφαρμογής. Μια διαφορετική δομή για τις εγγύσεις και μια διαφορετική δομή για τα δάνεια και την ε, ε, συμμετοχή. Συνολικά, μάλλον Παρά τις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίσαμε, μπορούμε με ιδιαίτερη χαρά να σας πούμε ότι οι μικροπιστώσεις λειτουργούν ήδη πλήρως. Επίσης, με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να σας πούμε ότι καταφέραμε να ετοιμάσουμε τη διευκόλυνση πολύ γρήγορα, πολύ αποτελεσματικά και πολύ συγκεκριμένα. Η οικονομική στήριξη της διευκόλυνσης ε, που θα είναι διαθέσιμη μέχρι το 2016, θα βοηθήσει τους ε, δικαιούχους μικροπιστώσεων και τους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς. Η μεγορά φυσικά εξελίσσεται, αναπτύσσεται και αυτό θέλουμε να το πετύχουμε φροντίζοντας να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, με την πανευρωπαϊκή προοπτική που έχουμε, πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πολύ καλή πρόσθετη αξία. Η πλατφόρμα τώρα κάλυψης που έχουμε για το Progress Microfinance θα βοηθήσει όλες τις μικροπιστωτικές μας πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ήδη δύο πειραματικέ δραστηριότητε, μία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μία άλλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ήδη υπήρξαν συνέργειες μεταξύ τους και πολύ καλά αποτελέσματα. Οι πέντε ενδιάμεση χρηματοδοτικοί φορεί που χρηματοδοτούνται βάσει της προπαρασκευαστικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνουν δικαιούχοι της Progress Microfinance πολύ σύντομα. Γι' αυτό και η Progress Microfinance έχει συνεισφέρει ήδη στη μεγαλύτερη συνοχή και στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ διαφόρων μικροπιστωτικών προγραμμάτων και μέσων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ζήτηση είναι μεγάλη και επανέρχεται ξανά και ξανά από την αγορά. Τα 100 εκατομμύρια προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρώθηκαν από αντίστοιχη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η δομή της διευκόλυνσης προβλέπει επίσης 47 εκατομμύρια επιπλέον πόρους από άλλους επενδυτές. Με τον καιρό και με τους διάφορους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς ελπίζουμε ότι το ποσό αυτό θα φτάσει στα 500 εκατομμύρια σε δάνεια για ατομικούς μικροδανιστές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, είμαι εδώ σήμερα για να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε με συγκεκριμένες δράσεις. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν πάρα πολύ. Τους τελευταίους μήνες, εκ με τη δημιουργία του μέσου αυτού διευκόλυνσης, έχουμε ετοιμάσει και συγκεκριμένες δράσεις. Επειδή ξεκινήσαμε νωρίς, μπορώ με ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα να σας πω ότι ήδη δύο υπογραφές για ε, επιχειρήσεις εγγυήσεων έχουν ε, προχωρήσει και είναι πολύ κοντά στο, στην ολοκλήρωσή τους. Πρόκειται είτε για μία επιχείρηση startup ε, MFI με μέλη διάφορους μη προνομιούχους από τις πόλεις και η δεύτερη περίπτωση είναι μια Ολλανδική ε, που αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση στις ε, συμβατικές αγορές επιστοτικών δανείων. Για τα δάνεια τώρα και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουμε 14 συγκεκριμένες δράσεις που βρίσκονται σε προθυμένο στάδιο προετοιμασίας και πιστεύουμε ότι το πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί για ένα ποσό που θα καλύψει ήδη την πρώτη παρτίδα πόρων και με τις εγγύσεις και με τα δάνεια κλπ. θα έχουμε συνεπώς 16 συγκεκριμένες δράσεις, 8 από τις οποίες είναι στην ε, Δυτική και 8 στην ε, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που έχουμε ξεκινάει αυτό το μέσο διευκόλυνσης. Οι συναλλαγές αυτές είναι επίσης και καλά ισορροπημένες. Το 1 τρίτο από αυτές γίνονται με τράπεζες και τα 2 τρίτα γίνονται με μη τράπεζες. Και για να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα για το πόσα πράγματα έχουμε καταφέρει, με τις δύο πρώτες ε, προσπάθειες εγγύησης υποβλήθηκαν για δάνεια και συμμετοχή στο κεφάλαιο και θα έχουν σαν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σε όργανα στην Ανατολική Ευρώπη ε, μικροπιστώσεων που θα βοηθήσουν ε, τον πληθυσμό των Ρώμα. Η δεύτερη περίπτωση είναι μια χρηματοδότηση για μια ομάδα μικρών οργανώσεων ε, ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα λοιπόν που ξεκινάει πλήρως η λειτουργία της διευκόλυνσης θα γίνουν προσπάθειες και στην αγορά γενικότερα με δίκτυα σε εθνικό επίπεδο με εκπροσώπησή μας σε, διάφορα, σε διάφορες εκδηλώσεις, με προσπάθεια ενημέρωσης και πρόθεσης του μέσου. Θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί φορείς της αγοράς. Ελπίζω με αυτά που σας είπα να καταλάβατε κάπως καλύτερα ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να ενημερωθήκατε και για τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας βοήθησε και μπορεί να θεωρηθεί ήδη μια επιτυχία κατά τη γνώμη μας. Βέβαια εννοείται ότι αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε με την επιτυχία αυτή σε όλο το στάδιο εφαρμογής της πιστοτικής αυτής διευκόλυνσης. Και ελπίζουμε να δείτε και εσείς τις επιπτώσεις και στις ε, αγορές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που λείπουν ε, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί όπως ε, ξέρετε έχουν και άλλα καθήκοντα να επιτελέσουν. Πολλά συμβαίνουν εδώ, πάντως ε, φανταζομαι ότι θα λάβουν και κάτι γραπτός από όλους σας, έτσι ώστε να το στείλουμε και σε όσους έπρεπε να επιστρέψουν στα κρατημέλη τους. Ε, Ήδη έχουμε στη διάθεσή μας ε, κάποια έγγραφα, αλλά αν θέλετε να προσθέσετε κι άλλα ε, στοιχεία θα τα στείλουμε στους βουλευτές που πρέπει να φύγουν λόγω καιρού. Από την Πολωνία είναι ο επόμενο ομιλητή και είναι εκτελεστικό διευθυντή ε, του Κέντρου Μικροχρηματοδότηση. Πρόκειται για τον κύριο Γκαλούσεκ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ εγώ εκπροσωπώ ένα δικτύο το οποίο είναι ενεργό στις χώρες ε, της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Συστήθηκε τη δεκαετία του 1990 και θέλω να πω λίγα λόγια για το πώς συστήθηκε το MFC, το Κέντρο Μικροχρηματοδότησης και πώς ε, έγινε ε, μέλος μιας οργάνωσης ήδη από τη δεκαετία του 90 γιατί μπορείτε ε, να ωφεληθείτε από τη λειτουργία του Progress και από την ανάπτυξη μηχανισμών μικροχρηματοδότησης εδώ στην Ευρώπη. Εμείς ως δίκτυο συστηθήκαμε λοιπόν το 97 όταν ε, οι κυβερνήσεις ε, ακόμη και οι τράπεζες ε, δεν θεωρούσαν ότι άξιζε να ξεκινήσουν τέτοια εγχειρήματα και εμείς ε, είχαμε κάποιους επιχειρηματίες που θέλουν να συστήσουν τις επιχειρήσεις τους, ε, αλλά δυσκολεύονταν ε, γιατί είχαν απολυθεί από κρατικές επιχειρήσεις, είχαν κρεοκοπήσει κάποιες επιχειρήσεις, όμως επρόκειτο για επιχειρηματίες που είχαν πάρα πολλές δεξιότητες και ήθελαν χρηματοδότηση για να μπορέσουν να στήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά. Έτσι λοιπόν αυτές οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες, στον Μπαγκλατές και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, προσαρμόστηκαν και στην Ανατολική Ευρώπη. Και τα προγράμματα τα οποία άρχισαν να λειτουργούν, έλαβαν επιχορηγήσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, λοιπόν, έλαβαν επιχορηγήσεις για 3-4 χρόνια και ε, είχαν κάποιους ε, θεσμικούς και προγραμματικούς στόχους ε, και αν, αν πετυχαίναν οι στόχοι τότε λάμβαναν δάνεια και για περαιτέρω ανάπτυξη και κατόπιν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην εμπορική χρηματοδότηση που σταδιακά θα ναι, γινόταν διαθέσιμη μέσω διάφορων ε, ιδρυμάτων που λειτουργούσαν παγκοσμίω. Δεν ήταν λοιπόν εύκολη διαδικασία, αλλά είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί τελικά να αποδείξουν την αξία τους στην αγορά. Και τώρα πώς έχει η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη μόνο έχουμε περίπου 60 διαφορετικούς οργανισμούς τέτοια ιδρύματα που ε, είναι βιώσιμα επιχειρησιακά μπορεί να καλύψουν το κόστος, δηλαδή το επιχειρησιακό κόστος ενώ όχι όλο το κόστος και ορισμένα αποδίδουν και κέρδος. Ε, και Τώρα, αν ε, κάνουμε ένα άλμα στο Progress, ε, παρά τα πολλά πλέον εκτήματα ε, για να έχουμε αυτή τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, τη δεκαετία 90 δεν θεωρούταν λογικό να αφιερώσουμε οποιαδήποτε χρηματοδότηση στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και δέκα έτη αργότερα υπάρχει αναγνώριση ότι η μικροχρηματοδότηση μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις startup ή τις υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις η υποδομή στην Ανατολική Ευρώπη ήταν αρκετά αδύναμη και εδώ βλέπουμε τις ε, γεωγραφικές διαιρέσεις και σε κάποιες από τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει μικροχρηματοδότηση και αναφέρομαι στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης μπορείτε να προσφέρετε ένα δάνειο ή μια εγγύηση, ενώ στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων. Τα περισσότερα προγράμματα δεν είναι βιώσιμα, τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι ακόμη και δύσκολο να πούμε ποιος οργάνωση είναι η κατάλληλη, ε, ποια ε, οργάνωση ασχολείται με τις startups, ε, ενώ ποιο ίδρυμα ασχολείται με άλλου είδους επιχειρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να οργανώσουμε αυτούς τους οργανισμούς με τη χρηματοδότηση. Δεν θέλω λοιπόν εδώ να υποσκάψω τη σημασία του progress, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας κρίκος που λείπει μεταξύ της ανάπτυξης αυτής της υποδομής που θα μπορούσε να απορροφήσει αυτή την ευκαιρία που έχουμε στη χρηματοδότηση του Progress. Ένα σημαντικό θέμα είναι το εξή, ότι η αναπτυγμένη έννοια τη μικροχρηματοδότηση είναι συμπληρωματική. Πάντοτε θα το λέω αυτό. Δεν ε, υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει τις υφιστάμενες δομές. Εδώ έχουμε πάρα πολλέ δομές μετοδότησης, έχουμε πιστοτικές ενώσεις, τράπεζες, Έχουμε ε, κάποια ιδρύματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις ε, μικρές επιχειρήσεις. Χρειάζονται απλώς ε, κάποια τεχνική βοήθεια και κάποια βούληση. Δηλαδή να υπάρχει βούληση της δίκησης να εργαστεί με αυτή την ομάδα και επίσης χρειάζεται τεχνική βοήθεια για να σχεδιαστούν τα σωστά προϊόντα. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στη μικροχρηματοδότηση και να σκεφτούμε, να λάβουμε υπόψη και τους υφιστάμενους ενδιάμεσους και να τους διευκολύνουμε στην δυνατότητα να ε, παράσχουν μικροχρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν το business model είναι σημαντικό, το επιχειρηματικό μοντέλο είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υφιστάμενες υποδομές ένα άλλο θέμα, το τρίτο θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω, έχει να κάνει με το εξής. Πολύ συχνά προσκρούμε στο ζήτημα της ικανότητας του πελάτη να απορροφήσει αυτή τη χρηματοδότηση, αυτούς τους πόρους. Δηλαδή έχουμε και ένα θέμα ε, χρήμα του οικονομικού αλφαβητισμού και υποστήριξης, ε, επιχειρηματικής υποστήριξης. Με το μηχανισμό Progress νομίζω ότι ε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υποδομές, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια και χρηματοδότηση για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής και την εξέλιξή της σε κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερο δυναμικό ως προς ε, την απορρόφηση της χρηματοδότησης Progress. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι από τη Γαλλία, είναι ο επικεφαλής της ε, μικροχρηματοδότησης ε, της ε, BNP, ο κύριος Τελούτσελ. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τον δικό μας μηχανισμό Γιασμίν και Τζέρεμι. Συμπληρώνονται από το δικό μας το μέσο. Σίγουρα μένουν πολλά ακόμα να κάνουμε και έχουμε και πολλά ακόμα να μάθουμε στην Ευρώπη για τα όσα συμβαίνουν στις χώρες του Νότου. Πριν να αναπτύξω τα διάφορα σημεία μου θέλω προηγουμένως να σας εξηγήσω που βρίσκεται η ΠΕΝΜΠΕ Παριμπά μέσα σε αυτόν τον μικρό κόσμο των μικροπιστώσεων. Πρόκειται για μια τράπεζα η οποία έχει κάποια πείρα στις μικροπιστώσεις και στις χώρες του Νότου αλλά και στις χώρες του Βορρά. Έχουμε εταιρική σχέση με το Λαντί που είναι ένας οργανισμός γαλλικός μικροπιστώσεων, ένας από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μπεν λοιπόν και η Παριμπά, από αυτές τις δύο φτιάχτηκε η Μπεν Παριμπά, εδώ και 17 χρόνια δουλεύουν για να δουλέψουν την Αντί και ως μεκίνες, δηλαδή τις δίνουν χρήματα για να αναπτυχθεί παρετέρω, αλλά και σε θελοντική βάση. Δηλαδή προσφέρουν τεχνική αρρωγή και προσφέρουν επίσης και θελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν τα διάφορα προγράμματά της. Ε, προηγουμένως, το είπε και ο κύριος Καλουτσά, δηλαδή αυτό που λέμε financial ε, literacy, δηλαδή πώς θα καταρτήσουμε και τους χρήστες, πώς θα μάθουν και αυτοί. Εδώ και 4,5 με 5 χρόνια ξεκινήσαμε μία δραστηριότητα η οποία συμπλήρωνε τις δραστηριότητες αυτές ε, που γίνονται σε θελοντική βάση και τις δραστηριότητες ε, χρηματοδότησης. Εγώ είμαι επικεφαλής του μικροπιστωτικού τμήματος με 300.000 δανειστές από τις νότιες χώρες. Δουλεύουμε με κάπου 20 οργανισμούς μικροχρηματοδότησης σε 10 περίπου χώρες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το κοινωνικό όφελος. Γνωρίζουμε ότι με τα 50 εκατομμύρια χρηματοδότησή μας φτάνουμε στο 80% περίπου γυναίκες. Το 80% είναι γυναίκες δηλαδή που υποφελούνται. Θέλουμε να στηρίξουμε παρετέρω την μικροχρηματοδότηση σε ολόκληρη όμως την Ευρώπη και όχι μόνο στη Γαλλία όπως γίνεται μέχρι τώρα. Και γι' αυτό αναπτύσσουμε, και ο τι θα αναφερθεί παρετέρω σε αυτό, γι' αυτό λοιπόν, όπως έλεγα, έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και με την Αντί στη Γαλλία, προκειμένου να δημιουργηθεί η εταιρική σχέση και με το Βέλγιο. Σε μερικές εβδομάδες θα έχει γίνει. Μικροστάρτ θα είναι το όνομά της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ε, συμμετέχει επίσης. Είναι δηλαδή μία από τις πρώτες προσπάθειες, αναπήραμα που κάνουμε για να συνεχίσουμε παρετέρω. Σας είπα λοιπόν ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύει η παριμπά για τις μικροπιστώσεις. Τώρα θα σας μεταφέρω και κάποιες σκέψεις μου για τις μικροπιστώσεις στην Ευρώπη σε σχέση με τις μικροπιστώσεις όπως αυτές λειτουργούν στον Νότο. Στην Ευρώπη είναι πολύ μικρές σε σχέσεις σε σχέση με τον Νότο. 150 εκατομμύρια έχουμε στον Νότο, ενώ λιγότερο από ένα εκατομμύριο δανειστές στο Βορρά σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροπιστώσεων. <clears throat> Για το κεφάλαιο 2% είναι η διαφορά. Βέβαια στο βορρά ε, το κεφάλαιο που ζητάνε είναι μεγαλύτερο. Πάντως, στο νότο σε σχέση με το παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Είμαστε όμως παρόλα αυτά πεπισμένοι ότι υπάρχει ανάγκη και ότι η ανάγκη αυτή ε, γίνεται ακόμα πιο μεγάλη δεδομένες της οικονομικής κρίσης που έχουμε σήμερα. Το ΕΦΕΗ πριν από μερικά χρόνια έκανε μία που κατέληξε στο ποσό των 700.000 ε, δανειστών, 7 δις δηλαδή, που θα χρειαστούν την υποστήριξή μας με μικροπιστώσεις. Εγώ πιστεύω ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί για να μην πω ότι θα τριπλασιαστεί διότι έχουμε 80 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν κάτω από τα όρια της ένδυας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό όπως καταλαβαίνετε και από αυτούς η μισή είναι οι φτωχοί εργαζόμενοι, δηλαδή άνθρωποι που έχουν δουλειά. Και μην ξεχνάμε ότι και οι άνεργοι είναι 10%. 24 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Άρα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, όπως και στην Ανατολική Ευρώπη μόλις έπεσε το τείχος του Βερολίνου, έτσι και σήμερα ακόμα και στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να έχουν μικροπιστώσεις. Δεδομένου βέβαια ότι τα χρήματα δεν είναι άπειρα, Πώς να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτή. Ίσως θα έπρεπε να εμπνευστούμε από αυτό που γίνεται στις χώρες του Νότου. Ήμουνα πριν από τρεις μέρες σε μια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Μικροπιστώσεων που έχει βάση στο Λουξεμβούργο αλλά που δουλεύει με χώρες του Νότου. 350 εμπειρογνώμονες από 80 διαφορετικές οργανώσεις ήμασταν εκεί. Και στο τέλος της ε, Εκδήλωση, ε, φτιάξαμε ένα ανακοινωθέν τύπου με τρία μηνύματα, τα οποία αποτελούν ακριβώς και τον τρόπο που θέλουμε να δουλεύουμε. Δηλαδή, η μικροπίστοση σήμερα στην Ινδία και στις χώρες γύρω από τον βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Η κατάσταση έχει μπλοκαριστεί εξαιτίας μέτρων τα οποία πήρε το κρατήριο του Μπραγκραντές που αρνείται νέα δάνεια και που κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη συλλογή των χρημάτων για την κάλυψή τους. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα μιλήσω για τα επιτόκια. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα δίχως άλλων στην Ευρώπη, λατινική θα έλεγα Ευρώπη, νότια Ευρώπη δηλαδή. Συχνά έχουμε δυσκολία να καταλάβουν πώς πληρώνεται ένα δάνειο ή πώς μπορεί κανείς να πληρώσει πάνω από 2% ή 5%. Πώς να ζητήσει δηλαδή κάποιος ένα τέτοιο επιτόκιο από τους φτωχούς δανειστές. Πριν όμως από 500 χρόνια έγινε ολόκληρη συζήτηση στην Καθολική Εκκλησία που είναι οι προκάτοχοι της μικροχρηματοδότησης. Υπήρχαν αυτοί που λέγανε πρέπει να δανείζουμε, α, μάλλον ότι το να δανείζουμε με ένα επιτόκιο, όποιο και αν είναι αυτό, είναι αμαρτία. Οι άλλοι, οι φραγισκανοί, λέγανε ότι μα πρέπει να καλύψουμε το κόστος του δανεισμού. Αυτή ήταν μια θεολογική συζήτηση λοιπόν, η οποία κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια. Τελικά αποφάσισε ο Πάπας με ένα κοσίλιο το οποίο ανέκρινε την απόφασή του αυτή και η απόφαση ήταν ότι πρέπει να καλύπτουμε το κόστος, άρα είναι απόλυτα θεμητό να βάζουμε ένα επιτόκιο, το οποίο όμως θα είναι λογικό επιτόκιο, έτσι ώστε, για να το πω με σημερινού όρους, να έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο που να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αυτό λοιπόν το παλιό δίλημα, το θεολογικό δίλημα, το ξαναβρίσκουμε και σήμερα στις χώρες του Νότου διότι ο μέσος όρος για την μικροχρηματοδότηση είναι 30% σήμερα ως επιτόκιο σε μερικές χώρες, μάλιστα φτάνει στο 80% και οι Μεξικάνοι λένε ε, κάτω από 55% δεν καλύπτουμε το κόστος. Είναι βέβαια συζητήσιμο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όσο πιο πολύ δανείζουμε, μάλλον όσο πιο μικρά δάνεια δίνουμε, τόσο μεγαλώνει το κόστος της ε, διανομής τους. Και τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος βέβαια επιστροφής. Είναι μια πραγματική συζήτηση αυτή. Μπορεί να υπάρχουν ε, λύσεις με συμπράξεις δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Πάντως, μικροχρηματοδότηση μπορεί να γίνει και να αναπτυχθεί με επιτόκια τη τάξη του 2%. Και αυτό που έλεγε ο Γκλουζέκ πριν από λίγο για το οικονομικό μοντέλο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δωρεάν δεν μπορεί να είναι. Κάποιο πρέπει να πληρώνει. Δεύτερον, εποπτεία, ρύθμιση και αυτορύθμιση. Στις χώρες του Νότου πολύ συχνά οι φορείς που προσφέρουν μικροχρηματοδότηση φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες, μια που δεν υπάρχει η κατάλληλη ρύθμιση για αυτούς. Αν δούμε και τη δουλειά που έχει κάνει η Αντί στη Γαλλία, που ήταν από τους πρώτους, κατάφερε να αλλάξει ο νομισματικός κώδικας, η νομοθεσία και έτσι επιτρέπεται μια εξαίρεση στο μονοπόλιο της τράπεζας να δανείζουν και πέτυχαν την άδεια να μπορούν να δανειστούν για να δανείσουν. Αυτέ είναι τροπολογίες πάρα πολύ σημαντικέ που έγιναν. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία, μην το υποτιμάμε. Η Επιτροπή τη Βασιλεία τώρα προχώρησε πριν από ένα χρόνο σε διαβούλευση με αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πριν από τρει μήνε. Ήταν για την εποπτεία και την ρύθμιση της μικροχρηματοδότησης. 52 σελίδε περίπου το έγγραφο αυτό και καταλήγει στο εξή. Επιμένει σε δύο πράγματα. Απ' τη μια ότι η ρύθμιση είναι σημαντικό να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση βέβαια για τις μικροπιστώσεις, συγχρόνως όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση. Το μήνυμα είναι έξυπνη ρύθμιση, καλά προσανατολισμένη στις ιδιωτερότητες της μικροχρηματοδότησης, που θυμίζει πάρα πολύ τις ε, ελληνικές τράπεζες. Στόχος είναι να βοηθάμε τους φτωχούς να αναπτύξουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Και γι' αυτό η περίπτωση της Γαλλίας είναι ιδιαίτερη. Έφτιαξε ένα παρατηρητήριο στα πλαίσια της Τράπεζας της Γαλλίας που να παρατηρεί ακριβώς τις μικροπιστώσεις. Στη Γαλλία λοιπόν μπήκαμε πολύ σε βάθος για να δούμε ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η μικροχρηματοδότηση. Δεν ξέρω κατά πόσο το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες, δεν νομίζω. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι μικροχρηματοδότηση και πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι πεπισμένος ότι η μικροχρηματοδότηση θα αναπτυχθεί μόνο εφόσον οι μικροί Ευρωπαίοι επενδυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή της. Σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό γίνεται αυτό, χάρη στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχουν ιστοσελίδες που φτάνουν μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες ή όπως το Babylon ή το Microworld στη Γαλλία που επιτρέπουν να δανείζει κάποιος μικροεπενδυτής σε έναν χρηματοδοτικό φορέα 20 ευρώ για παράδειγμα, από 20 ευρώ και πάνω. Στην περίπτωση της Γαλλίας υπάρχει ρύθμιση και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Είναι μια δυνατότητα λοιπόν που υπάρχει για τους Ευρωπαίους πολίτες χάρη στο διαδίκτυο. Με ξέρεις όμως κάποιες χώρες όπως είναι το Λουξεμβούργο και κάτω χώρες, κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι μικρές τράπεζες δεν μπορούν ε, να δώσουν ε, χρήματα για μικροπιστώσεις στους πελάτες τους. Είναι κάπως παράδοξη κατάσταση αυτή, γιατί η ζήτηση υπάρχει. Οι πελάτες θα θέλανε. Γιατί να μπορούν να το κάνουν μόνο στο Λουξεμβούργο και στις κάτω χώρες. Οι τράπεζες όμως δεν μπορούν να δώσουν τέτοια ε, χρήματα διότι οι ρυθμιστές τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο δεν τους το επιτρέπει. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι τέτοιου είδους πιστώσεις, αν δούμε το κίνδυνο και τις κοινωνικές επιπτώσεις, θα έπρεπε να επιτρέπονται, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες παρατηρήσεις μου για να καταλάβετε πώς έχει η Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, τι θα γίνει. με το Progress. Έξι δις πιστώσεις, 700.000 ε, δανειστές, έχει ξεπεραστεί βέβαια ήδη αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη, πραγματική ζήτηση. Η κάλυψη του κόστους τώρα των ε, μικροπιστωτικών ιδρυμάτων δεν αποδίδουν, εννοείται. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ποσό που να είναι σε θέση να φτάσουν σε ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί έτσι θα γίνει το ντεκλίκ και θα μπορέσουν να αποδώσουν περισσότερο. Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, πρέπει οι ρυθμιστές να καταλάβουν ποια είναι η ιδιαιτερότητα της μικροχρηματοδότησης. Όχι μόνο την οικονομική, δημοσιονομική πτυχή, αλλά να δουν λιγάκι και την κοινωνική πτυχή. Και θέλω εδώ να επιμείνω για το ότι πρέπει να αποφύγουμε την ψευδέστηση ότι με την μικροχρηματοδότηση θα απαλείψουμε την ε, φτώχεια. Πριν από 50 χρόνια με το βραβείο Νόμπελ είδαμε ότι υπήρξε μεγάλο ενθουσιασμός. Σήμερα όμως είναι σε κρίση όπως σας είπα οι Τι θέλει, υπό λοιπόν αμφισβήτηση. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία του παρελθόντος. η μικροχρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο μπορεί να βοηθήσει, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να χτίσουμε ένα οικονομικό μοντέλο που να είναι ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο να στέκει στα πόδια του. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλο ένα θέμα πριν το μεσημέρι, διότι είχαμε μια αλλαγή στην ημερησία διάταξη λόγω του καιρού. Επόμενος ομιλητής είναι από την Ουγγαρία, είναι διευθυντής ε, της ε, πρωτοβουλίας ε, μικροχρηματοδότησης, ο κύριος Ουσλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ε, δεν το σκόπευα, αλλά νομίζω ότι θα έχω μια συζήτηση με τον διπλανό μου. αλλά η πρώτη μου πρόταση είναι ότι στην παρουσίαση αυτή θα ήθελα να ε, υπερασπιστώ ένα MFI για να ε, διευρύνουμε τις δυνατότητες μικροχρηματοδότησης ε, σε φτωχούς Ρώμα, παρότι ένα τέτοιο μηχανισμός δεν πρόκειται να είναι επικερδής, δεν θα είναι δηλαδή βιώσιμος. Ή, εν μέχρι ένα βαθμό μόνο. Το ερώτημα είναι αν ε, μπορούμε να αντιγράψουμε ένα τέτοιο μηχανισμό και αν αξίζει να τον μιμηθούμε. Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Η εμπειρία μου στο θέμα αυτό προέρχεται από τη συμμετοχή μου στον σχεδιασμό του ε, Ουγγρικού MFI που λέγεται CUTE Program. Το ...ο οποίο χρηματοδοτείται από το πιλωτικό πρόγραμμα για τους Ρώμα της Γενικής Διεύθυντης για τις Περιφέρειες. Ε, μάλλον θα γνωρίζετε αυτό το πειραματικό πρόγραμμα. Ε, έχουμε λοιπόν ε, το πιλωτικό πρόγραμμα για τους Ρώμα και είναι πολύ σημαντικό μέσω αυτό για το κίνημα κοινωνικής ένταξης των Ρώμα στην Ανατολική Ευρώπη αποστολή του προγράμματος ε, είναι να βοηθήσει ε, φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, κυρίως Ρώμα, να βελτιώσουν ε, με αξιοπρέπεια την κατάστασή τους, παρέχοντάς τους χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πληροφόρηση και κοινωνική βοήθεια. Αυτό δηλαδή μοιάζει πολύ με αυτά για τα οποία μιλήσατε εσείς. Θα ήθελα να σας περιγράψω πρώτα ποιοι είναι οι Ρώμα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα εκτός της Ευρώπης ε, Κανείς ε, δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι Ρώμα. Πιστεύουν ότι είναι μια μικρή μειονότητα που φοράει πολύ χρωμαρούχα και τους αρέσει να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αλλά στην πραγματικότητα, στην Ανατολική Ευρώπη, η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το συζητάμε. Στην Ουγγαρία ε, αποτελούν περίπου το 7 ή 8% του πληθυσμού. Ε, μιλάμε δηλαδή για σχεδόν το 1 εκατομμύριο ένα εκατομμύριο είναι αυτοί που, που έχουν χάσει περισσότερα ε, από την αλλαγή καθεστώτος του 1990, διότι το κομμουνιστικό καθεστώς είχε μια πολύ κακοσχεδιασμένη πολιτική ένταξη έκανε τους Ρώμα να εργάζονται στην βαριά βιομηχανία, να κάνουν τις ανειδίκευτες εργασίες ε, και στα στις εκμεταλλεύσεις των συνεταιρισμών. Μόλις ιδιωτικοποιήθηκαν τα πράγματα, ε, όλη τη δουλειά τους. Ε, υπάρχει λοιπόν ποσοστό ανεργίας σε 35% για τους άνδρες και 20% για τις γυναίκες ε, που είναι μάλλον το χειρότερο ποσοστό ανεργίας που έχουμε δει. Αυτό εντείνεται από τον κοινωνικό αποκλεισμό την καταστροφή των παραδόσεών τους που δεν μπορεί να διατηρήσει κανείς όταν δουλεύει στη βαριά βιομηχανία. Ε, υπάρχει απομόνωση στα γκέτο, ε, σχολεία όπου υπάρχει διαχωρισμός. Ε, ε, πολύ λίγα παιδιά προχωράνε στο Λύκειο. Το 10% των Ρώμα ε, συμμετέχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τον υπόλοιπο πληθυσμό το ποσοστό είναι 80%. Και ένα τελευταίο νούμερο για τους Ρώμα, το 70% έχει εισόδημα που βρίσκεται στο τελευταίο πέμπτο του πληθυσμού, στο τελευταίο 20%. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να βρούμε ένα μέσο για τους Ρώμα. Οι κυβερνήσεις μας τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά έχουν ε, εισάγει κάποια ωφέλη, κάποια ε, επίδομα ανεργίας ε, και κάποια άλλα κοινωνικά επιδοτήματα που δεν είχαμε την κομμουνιστική εποχή, αλλά πέρα από, αυτά τα, πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις δεν είχαν καμιά καλή ιδέα για το πώς να λύσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό με κάποιους φίλους προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι. Διαβάσαμε λοιπόν το φημισμένο βιβλίο και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Ε, ένας από τους διευθυντές της ε, Ράιφ Άιζεν ε, συμμετέχει. Ε, είχε βοήθεια από ε, ανώτερα στελέχη της Deloitte Λετούς ε, και άλλους. Το ξεκινήσαμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό με δικά μας χρήματα και ε, σαν μάνα εξ ουρανού ήρθε η Γενική Διευθυνσή Ρέτζιο και μας έδωσαν κάποια χρήματα. Ουσιαστικά θέλαμε δάνεια χωρίς εγγυήσεις τα οποία δεν είναι πολύ εύκολα σύμφωνα με τον κανονισμό. Μιλάμε για μικρά ε, ποσά. Το μεγαλύτερο ποσό είναι 3.500 ευρώ. Στοχεύουμε κυρίως στους ανέργους, ε, τους ε, ανεκπαίδευτους Ρώμα. Ο στόχος είναι μόνο για την δημιουργία εισοδήματο. Δεν δανείζουμε λοιπόν για στέγαση και τέτοια. Είναι ένα πρόγραμμα δανεισμού προς ομάδες. Ε, θέλουμε να συμμετέχουν 4 με 7 άτομα στις ομάδες ε, και ε, υπάρχει η πίεση των ομοτήμων αντί για εγγύηση. Επίσης, ο δανεισμός γίνεται διαδοχικά, δηλαδή πρώτα δύο μέλη της ομάδας λαμβάνουν χρήματα. Όταν αρχίσουν αυτοί να επιστρέφουν το δάνειο, τότε προχωράμε. Η πληρωμή των δόσεων γίνεται εβδομαδιαίως ενθαρρύνουμε την αποταμίευση και έχουμε 10% περιθώριο ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού και τα επιτόκια καταθέσεων. Η Ουγγαρία είναι δύσκολη χώρα διότι προφανώς ο καθένας πιστεύει ότι η χώρα του είναι δύσκολη αλλά εμείς το νιώθουμε ε, διότι υπάρχει υπερβολική ρύθμιση και ε, σημαντική γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, μια τράπεζα δεν ενδιαφέρεται να, ε, κάνει, να, να μπει στον τομέα του κοινωνικού μικροδανισμού. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα MFI, να μην μπω σε λεπτομέρειε, αλλά αποφασίσαμε να έχουμε διτή δομή. Έχουμε από τη μία την εμπορική τράπεζα, Raiffeisen, και από την άλλη έχουμε το MFI, το οποίο είναι ξεχωριστό. Το μέσο μικροχρηματοδότησης δηλαδή. Η τράπεζα χρηματοδοτεί και ε, χειρίζεται τον μηχανισμό αυτό. Ε, ζητήσαμε από την ε, κυβέρνηση να εγγυηθεί για τα δάνεια, αλλά αυτό δεν έγινε. Η Ράιφ παρέχει 400 εκατομμύρια. Έχουμε συνολικά δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, το περιθώριο 10% ανάμεσα στα επιτόκια ε, στόχο έχει να καλύψει τις απώλειες. Ε, Πολλέ υπηρεσίε είναι δωρεάν για του πελάτε μα και τελείω ξεχωριστή οντότητα είναι το MFI. Εμεί απασχολούμε τους ανθρώπου που εργάζονται πρακτικά με τα ζητήματα αυτά, που κάνουν τι πρακτικέ έρευνε. Δεν πιστεύουμε ποτέ ότι θα έχουμε κέρδος από αυτό. Ακόμα και αν έχουμε 20.000, 30.000 ή ακόμα περισσότερους πελάτες, ποτέ δεν θα έχουμε κέρδος. Ούτε καν στοχεύουμε να έχουμε κελισμένους ισολογισμούς. Ε, αλλά όλοι, ο, ο, ο, ε, είναι διευθυντής της τράπεζας, οπότε βγάζει κέρδος από εκεί. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο ε, δανείων εκ των οποίων μόνο το 10-15% να πηγαίνει στους Ρώμα για να ε, λέμε ότι κάνουμε καλό. Είναι μια κοινωνική ε, προσπάθεια. Μας ενδιαφέρει ο κοινωνικός αντίκτυπος. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε και στα νούμερα να το δούμε αυτό, διότι έχουμε, έχουμε το κόστος ενός δανείου. Θα το δούμε αυτό στο τέλος του πειράματος που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή. Εάν το κόστος αυτό είναι μικρότερο από, την, ε, από τα ωφέλη που λαμβάνει μία άνεργη οικογένεια, αν είναι χαμηλότερο δηλαδή από το επίδομα ανεργίας που θα λαμβάνει μια ανεργή οικογένεια, τότε νομίζω ότι θα μπορούμε να υπολογίσουμε ποιο είναι το κόστος και πώς αντισταθμίζεται από τον κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος. ε, λάβαμε μια σοβαρή απόφαση που μπορεί να ακούγεται πολύ δραματική, ε, μπορεί να ακούγεται λιγότερο δραματική σε άλλες χώρες από ότι στην Ουγγαρία. Αποφασίσαμε να χρηματοδοτούμε μόνο νόμιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει δηλαδή να καταχωρούνται ε, οι, ε, αυτοί που λαμβάνουν δάνεια. Αυτό είναι ε, σημαντικό επιπλέον διοικητικό άχθος. Αποφασίσαμε όμως ότι δεν θέλουμε να χρηματοδοτούμε ανθρώπους στην μαύρη αγορά. Κάποιες άλλες χώρες το κάνουν αυτό, ιδιαίτερα για τους ε, Ρώμα, η Ρουμανία, η Μακεδονία λέει ο μιλητής, ε, αλλά εάν δεν μπορέσουμε να του εντάξουμε στον κανονικό επιχειρηματικό κόσμο θα είναι άχρηστο αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε διαφανείς επιχειρήσεις. Ένας άνεργος ε, Ρώμα λαμβάνει 100 ευρώ το μήνα ως ε, κοινωνικό επίδομα και υποτίθεται ότι η οικογένεια ζει από αυτό. Αλλά από τη στιγμή που θα ε, καταχωρηθεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας η κυβέρνηση θεωρεί ότι ε, εισπράττει το ελάχιστο εισόδημα που είναι, 400, είναι 300 ευρώ το ε, μήνα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αρχίσει να πληρώνει κοινωνικές αποδοχές ε, να πληρώνει και κοινωνικέ εισφορέ. Ήδη από την πρώτη μέρα δηλαδή, που δεν έχει, όχι κέρδο, δεν έχει ούτε τζίρο, ο άνθρωπο αυτό χρεώνεται. Εάν θέλει να καταχωρηθεί ως ε, ε, ε, έμπορος που μετακινείται από τόπο σε τόπο, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να περάσει πρώτα εξετάσεις. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να μελετήσει 70 ώρες μεταξύ άλλων αγγλικά. Φανταστείτε τώρα μια γυναίκα Ρώμα που ούτως ή άλλως πουλάει λαχανικά για να μπορεί να καταχωρηθεί ως ελεύθερος επαγγελματία και να πληρώσει τις κοινωνικές φορές, θα πρέπει να περάσει εξετάσεις αυτές που στοιχίζουν και χρήματα και θα πρέπει να μάθει ε, να μιλάει ε, ε, επιχειρηματικά αγγλικά. Τι να τα κάνει αυτά στο, στον υπόγειο, στο σταθμό του υπογείου που θα δουλεύει. Εμείς εργαζόμαστε ως εξής εντοπίζουμε κάποια σημαντικά γκέτο των Ρώμα και σε χωριά και σε πόλεις. Οι εργαζόμενοι μας ε, πηγαίνουν εκεί, δεν ρωτάνε τον κόσμο αν είναι Ρώμα ή όχι. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιο ε, που είναι εκεί ε, είναι Ρώμα. Αν δεν είναι και πάλι ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει. Προσπαθεί λοιπόν να εντοπίσει τις ομάδες για να υπάρχει συνοχή μεταξύ των ανθρώπων. Έχει ε, συναντήσεις μαζί τους. Ε, στην αρχή, η αρχή είναι πάντα δύσκολη, διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τελικά προχωρούν. Ε, στόχος ήταν να συνδυάσουμε ε, αυτήν την κοινωνική προσπάθεια ε, με ένα λογικό επίπεδο επιχειρηματικών συμβούλων, διότι κάποια στιγμή καταλήγει η συζήτηση στο τι, τι επιχείρηση θα θέλετε να δημιουργήσετε, πώς θέλετε να βγάλετε χρήματα και πώς πιστεύετε εσείς ότι θα λειτουργήσει αυτό. Είσαστε βέβαιο ότι θα μπορέσετε να ε, πληρώσετε το δάνειο. Είσαστε σίγουροι ότι θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό σε εβδομαδιαία βάση. Ε, προχωρούν λοιπόν ε, στα θέματα λογιστικής, προχωρούν σε συμβουλές σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, εάν ε, χρειαστεί να αγοράσει ο άνθρωπος το αυτοκίνητο. Ε, είναι λοιπόν ένα θέμα επιχειρηματικών ε, συμβουλών που δεν έχουν δει ποτέ οι πελάτες μας στο παρελθόν, διότι έχουμε δει και άλλα προγράμματα μικροχρηματοδότησης ε, εάν έρχεται λοιπόν κάποιο, ε, λέει θέλω χειροστάσιο, ε, του δίνουν τα λεφτά, μετά από κάποιου μήνε μήνες ε, ξαναπερνάει από εκεί ε, ο δανειστής και μπορεί να, μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος, μπορεί, μπορεί όχι. έχουμε λοιπόν θέσει κάποια κριτήρια επιτυχίας για μας. Λέμε ότι εάν δεν εξυπηρετούνται το 70 ή 80% των δανείων, τότε δεν προτείνουμε εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Ξέρετε τα στοιχεία της ε, Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ποτέ το 95%. Ε, εάν όμως ε, πληρώνεται το 70% των δανείων, τότε το 10% το πληρώνει η τράπεζα και Έχουμε και 10% περιθώριο. Θέλουμε επίσης ε, οι ε, πελάτες μας που πληρώνουν το δάνειο τους ε, να λάβουν ένα δεύτερο δάνειο το οποίο δείχνει ότι τουλάχιστον η επιχείρησή τους τρέχει. Και θέλουμε να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο. Υπολογίζουμε λοιπόν πόσο στοιχίζει ένα δάνειο και πόσο και πόσο εισόδημα έχουν οι άνθρωποι αυτοί θεωρητικά για το, σύμφωνα με το κράτος. Η Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειών έχει δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης ε, της ε, συνέχειας. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το UNDPR παρακολουθούν τις προσπάθειές μας ε, θα ήθελα να πω το εξή, ότι είναι πολύ αισιόδοξο το να πηγαίνει κανείς ε, στα χωριά αυτά, διότι ο κόσμος ε, κανονικά ζει πίσω από κλειστές πόρτες, ε, ανησυχεί σχετικά με τις συνθήκες, πώς να επιβιώσει κανείς με 100 ευρώ το μήνα, αναζητούν νόμιμη εργασία, οι εργοδότες τους ξεγελάνε, τους εξαπατούν. Ε, με, με τη δουλειά μας όμως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Ο κόσμος αρχίζει και ευχαριστιέται τις εβδομαδιαίες εβδομάδες, αρχίζει γνωρίζεται μεταξύ τους. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτές τις μικρές ε, κοινωνίες ε, πολλοί ε, κόσμος γελάει με τους ανθρώπους που έρχονται στις συναντήσεις που οργανώνουμε. Τους λένε ότι α, και αυτοί θα, θα, σας, θα σας εξαπατήσουν, θέλουν τα χρήματά σας, θέλουν την κόρη σα. Ε, αλλά οι άνθρωποι που πραγματικά συνέχισαν να έρχονται στις ε, συναντήσεις αυτές και έλαβαν τα πρώτα δάνεια, είδαν ότι μπορούν να πάνε να αγοράσουν πράγματα που θέλουν. Κάποιους από αυτούς τους δίρανε, διότι αμέσως ήρθαν, ήρθε η οικογένεια και έλεγε ότι «Α, έχεις χρήματα, μπορείς να μου δανείσεις». Ενώ αυτοί οι άνθρωποι αρνηθήκαν να δανείσουν τα χρήματα που είχαν λάβει. Ε, θα επιδείξω κάποια σημεία διότι έχω μακρηγορήσει. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν μπορεί να αναμένει κανείς ε, ένας τέτοιος μηχανισμός να, ε, ε, να παράγει κέρδος. Όχι με τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε εμείς και με το, τους στοχευμένους πελάτες που έχουμε. Ε, πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί να δημιουργήσει μια δομή, ένα μηχανισμό όπου να ε, χρηματοδοτείται, ε, όπου να μην υπάρχει αρχική χρηματοδότηση, αλλά όπου να υπάρχει ενίσχυση της ε, λειτουργίας. Νομίζω ότι οι τράπεζες θα θέλουν να το κάνουν αυτό, δεν ε, θέλουν όμω να κάνουν να κάνουν όλη τη δουλειά, διότι δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή. Τα, το κόστος λειτουργίας θα πρέπει να καλυφθεί και αυτό είναι ακριβό. Ελπίζουμε η ε, Παγκόσμια Τράπεζα και η UNDP να ε, μας στηρίξει και να έχουμε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελικός ομιλητής ε, του να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις είναι ο Γενικός Διευθυντής της Microstart, ο κύριος Σαπί. Δέκα λεπτά έχετε. Αν μπορείτε να περιοριστείτε στα δέκα λεπτά θα είναι χρήσιμο. Θα προσπαθήσω, θα μιλήσω γαλλικά εκπρόσωπο την κυρία Νόβακ, η οποία δυστυχώς για λόγους υγείας πρέπει να στο Παρίσι και μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω εδώ. Ε, πριν να προσεγγίσω την ουσία του ζητήματος, να σας αναφέρω ποιο είναι το πλαίσιο σχετικά με τη μικροπίστωση στην Ευρώπη. Εδώ και 20 χρόνια η μικροπίστωση γνωρίζει σημαντική άνθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες η λογική είναι εξής, ανάπτυξη των υπηρεσιών που σε ορισμένα κράτη συνοδεύτηκε σε μια επιταχυνόμενη αποβιομηχανοποίηση, αύξηση της ανεξάρτητης εργασίας και δυστυχώς οικονομικές κρίσεις ε, που καταρχήν ε, πλήττουν τους ε, πλέον ευάλωτους. Αυτά είναι στοιχεία που συνεισφέραν στην ανάπτυξη της μικροπιστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προσθέσουμε, όπως είπε ο κ. Ζέλ προηγουμένως, ε, ε, ένα ενδιαφέρον και μια συμμετοχή αυξανόμενη των εμπορικών ε, τραπεζών που βλέπουν μια δυναμική στην αγορά ή μια δυνατότητα να παγιώσουν την εταιρική τους ευθύνη με δράσεις που αφορούν την καρδιά του, του κλάδου τους αλλά και των κρατών και των ευρωπαϊκών οργάνων και των ευρωπαϊκών χασμών. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν θεσπίσει μια σειρά καινοτόμων εργαλείων που επέτρεψαν σε ε, δεκάδες μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης να αναπτυχθούν. Δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας το 2007 ε, ε, έχουμε τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης και ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, έδωσαν μια σημαντική χρηματοδότηση. Ε, έχουμε και το Jasmine, το εργαλείο τεχνικής βοήθειας που ξεκίνησε το 2009. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι μηχανισμοί και τα γνωρίζω αυτό που σας λέω, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να βελτιώσουμε το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της μικροπίστησης και των μικρών επιχειρήσεων. Υπάρχει μία σειρά εμποδίων για την ανάπτυξη της μικροπίστωσης που πρέπει να αρθούν φυσικά στα κρατη Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη συστήσει ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια που μπορούν να επιτρέψουν να αναπτύξουν μικροπιστό στην Ευρώπη. Αφενός, ε, σε ό,τι αφορά την ε, ε, χρηματοδοτική ρύθμιση. Έχουμε ε, και τα δύο παραδείγματα. Έχουμε ε, την αφαίρεση των ατοτοαρίου του ρυθμού απομειώσεων που αφορά τη δυνατότητα δανεισμού και των μικρών δανείων και τη δυνατότητα δανεισμού για νέο δανεισμό. Αυτά σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία αλλά δεν ε, υπάρχει επίσης ούτε εναρμονική ανάπτυξη των ε, ε, καθεστώτων για, τις, για τα ελεύθερα επαγγέλματα στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης. Ε, όμως η θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών ε, επιτρέπει από το 2007 να έχουμε πάρα πολύ σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη. Ε, αναπτύχθηκαν παντού μηχανισμοί μικροχρηματοδότηση στην Ευρώπη, το Jasmine και το Progress επιτρέπουν στους οργανισμούς μικροπίστωσης να εγγυθούν ότι τα χαρτοφυλακιά τους λαμβάνουν ε, ενδιαφέροντα επιτόκια και να αποκτήσουν ε, μία μορφή σε ίδια κεφάλαια με τη μορφή κεφαλαίου καθώς και να αποφεληθούν τεχνικής βοήθειας, κάτι που είναι απαραίτητο για τους μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης. Ε, τώρα, οι πιο συγκεκριμένα παραδείγματα που είναι και πιο κοντά σε εμά που μπορούμε να δούμε για να σας δείξουμε το Βελινικές ε, είναι η, πρόσφατη σύσταση της ε, ε, συνεταιριστικής εταιρείας Microstract με κοινωνικούς στόχους η οποία ε, στην οποία συμμετέχει η Μπεν Πέπα ε, Φορτής ε, στο Βέλγιο και ελπίζω και σύντομα να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η Μικροστάτ δημιουργήθηκε μεταξύ συνεργασίας του Άντι και της BNP Paribas στο 2010 αποφάσισαν οι εταίροι να δημιουργήσουν έναν οργανισμό μικροπίστωσης που θα πρέπει να υποδεχτεί τους πρώτους του πελάτες τον Ιανουάριο του 2011 εδώ στις Βρυξέλλες. Σε αυτό το πιλωτικό σχέδιο, το οποίο λειτουργεί σε δύο συνοικίες ε, των Βρυξελών, το αρχικό κεφάλαιο, ε, το προσφέρει BNP Paribas Fortis και ε, ελπίζω να συμμετάσχει σύντομα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η Άντι ε, συνεισφέρει με την εμπειρογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία. Η ΜΠΕ Περιβά πέρα από το κεφάλαιο ενεργοποιεί πιστώσει 750 εκατομμυρίων προκειμένου να μπορεί η μικρόστρατη να χρηματοδοτήσει με επιτόκια τη αγοράς και το ε, ΕΤΕΠ ε, εγγυάται συμμετοχή γύρω στο 75% ε, και ελπίζουμε ότι από το Δεκέμβριο του 2010 θα συμμετέσχει. Η Άντι Μπέρν και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ισχύουν τη συνεργασία τους μέσω της ε, Microstat και δημιουργούν κάτι μοναδικό στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια δημόσια, εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού στομέα, ιδιαίτερα καινοτόμη που θα χρηματοδοτήσει και θα συνοδεύσει 800 νέους πελάτες στην πιλωτική φάση αυτή που θα διαρκέσει στο 2012. Ένας ε, από τους στόχους ε, που θέλουμε να πετύχουμε είναι να καταδείξουμε ότι το ε, οικονομικό μοντέλο του Μικρόστρατε θα μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί από το 2017 και επομένως θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιβίωσή του μακροπρόθεσμα. Αυτό φυσικά για το καλό των πελατών. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω ε, κάποιες πτυχές γιατί αν μπορέσει να συνεχίσει να αναπτύσσεται η μικροπίστωση στην Ευρώπη ε, θεωρούμε ότι έχουμε τρία ε, θέματα που διακυβεύονται και που πρέπει να εντοπίσουμε. Καταρχήν ε, η υλοποίηση ε, από τα ευρωπαϊκά όργανα προγράμματα στήριξης προσερμοσμένα για τους ε, μικρούς μηχανισμούς μικροχρηματοδότησης τα εφιστάμενα μέσα έχουν επιτρέψει στους μηχανισμούς να αναπτυχθούν σημαντικά παρόλα αυτά για τη δημιουργία μικρών τέτοιων οργανισμών μικροπίστωσης ε, που έχουν δυσκολίες ε, να διαχειριστούν το επίπεδο πολυπλοκότητας ε, των μηχανισμών και να αναπτύξουν συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Το δανεικό θα ήταν να θεσπιστεί ένα σύνολο απλοποιημένων υπηρεσιών υπό τη μορφή πακέτου για τις, τους μικρούς μηχανισμούς χρηματοδοτήσεις θα μπορούσαμε εδώ να μιλάμε για ε, εγγυήσει ή πιστώσει, ε, δηλαδή χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και μια μικρή επιδότηση ε, που θα δίνεται στην αρχή για την εκκίνηση και δεν θα, ε, δεν θα πληρώνεται πίσω. Επίσης θα έπρεπε με κατάλληλο τρόπο να δεσμευτεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στη βάση ενός business plan. Δεύτερον, στο πλαίσιο του Single Market Act και της προετοιμασίας του Bond Business Act θα πρέπει ε, να ε, προωθηθεί η ανάπτυξη της μικροχρηματοδότησης. Ε, η ανάπτυξη μικρών παραγωγικών μονάδων ανεξάρτητων στην Ευρώπη είναι μια τάση που θα επιταχυνθεί στη Γαλλία από το 2009 η υλοποίηση του καθεστώτος του ανεξάρτητου επιχειρηματία οδήγησε στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων γιατί ε, πολλά φορολογικά και κοινωνικά εμπόδια είχαν αρθεί για τις ε, μικρές επιχειρήσεις ένα ευρωπαϊκό ε, καθεστώς ε, του ανεξάρτητου επαγγελματία θα μπορούσε να δει το φως τα επόμενα χρόνια και αυτό φυσικά ε, θα ενθάρρυνε τις εξελίξεις αυτές. Ε, επίσης, ε, τα εμπόδια εισόδου στις μικρές δραστηριότητες θα μπορούσαν να έρθουν πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν θα διευκολύναμε την πρόσβαση των νέων και των λιγότερο εξειδικευμένων σε αυτά τα εγχειρήματα. Το τρίτο θέμα που διακυβεύεται αφορά μία πρόταση σε σχέση με ένα ε, πλαίσιο που να ευνοεί περισσότερο το τη μικροχρηματοδότηση, η ανάπτυξη ε, Τη ε, εταιρική επιχειρηματικότητα, Social Coalition στην Αγγλία, Positive Entrepreneur στο Βέλγιο, ε, μας δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό κίνημα η περιοχή του κοινωνικού σκοπού έναντι τη άμεση αναζήτηση κέρδου, το επιχειρηματικό πνεύμα ή σύσταση οικονομικών μοντέλων βιώσιμων ε, ε, ε ιδιωτικής και δημόσιας, με πόρου ιδιωτική και δημόσιας προέλευσης είναι αρκετοί δείκτες που ε, στηρίζουν ε, τους μηχανισμούς μικροχρεοδότησης. Ε, η σύσταση ενός ευρωπαϊκού καταστατικού ή μιας εταιρείας με κοινωνικούς σκοπούς θα μπορούσε να ευνοήσει στην αναγνώριση των μηχανισμών μικροχρηματοδότησης που υπάρχουν στην Ευρώπη και θα μπορούσαμε να προβούμε και σε μια σύγκριση των μοντέλων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα εργαλείο που να εξυπηρετεί και τις μικρές επιχειρήσεις ε, και ε, τους πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία. Μιλάμε για ένα μέσο οικονομικού δημοκρατισμού, που θα μπορούσε να επιτρέψει στους πολίτες να λάβουν οι ίδιοι τη μοίρα τους στα χέρια τους. Πρόκειται για ένα εργαλείο ε, κοινωνικό ευρωπαϊκού συνδέσμου που συνεισφέρει στην κοινωνική συνοχή της Ευρώπης και που συνεισφέρει στο να αποκτήσει δυναμική η Ευρώπη έναντι της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο σας. Θα ήθελα να τελειώσουμε την ακρόαση αυτή μέχρι τις 12, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας για τους Ρώμα. Όμως, προηγουμένως, κατάλογος ομιλητών. Η κυρία Ζαζοφιέσκα είναι η πρώτη που έχει ζητήσει το λόγο για να υποβάλει ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια που καταφέραμε και είχαμε τόσο υψηλό επίπεδο πυρογνώμονε στην ακρόασή μα. Χαίρομαι πραγματικά γιατί επιστρέφουμε σε μια καλή παλιά παράδοση που είχαμε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σας, ειλικρινά. Ακούσαμε για το βαθμό εφαρμογής από την κυρία Μπρουν Λεόν του μικροπιστωτικού μέσου. Πόσα χρήματα χρειάζονται για μια startup επιχείρηση, για μια μικροεπιχείρηση, ιδιαίτερα μικρή επιχείρηση. Με εκπλήσει όμως το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Υπάρχει κάποιος λόγος, δεν είναι καλά ενημερωμένες ε, οι επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν ε, οι μικροπιστώσεις αυτές να φτάσουν ε, στους δικαιούχους τους. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί. Είπατε επίσης ότι στην Ανατολική Ευρώπη τα χρήματα πηγαίνουν κυρίως για να στηριχθούν οι Ρώμα, ενώ στη Δυτική Ευρώπη πηγαίνουν κυρίως για να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό με απασχολεί κάπω. Δεν είναι ότι δεν είμαι υπέρ των Ρώμα. Έρχομαι από μια περιοχή η οποία έχει μια πολύ μεγάλη γερμανική μειονότητα και μειονότητα των Ρώμα. Θεωρούμε ότι είμαστε πολυπολιτισμικοί και ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις εθνικές μειονότητες. Η δουλειά που γίνεται με τους Ρώμα είναι πολύ καλή. Είναι για μας, θεωρούμαστε μάλλον μοντέλο για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα ζήτημα των Ρώμα. Ο κύριος ε, Ντελούτσελ είπε ότι θα μπορούσαν να τεπλασιαστούν τα ποσά, γιατί υπάρχει ανάγκη. Συγχρόνως όμως τόνισε ότι τα μικροδάνεια είναι μια διευκόλυνση υψηλού κινδύνου που εξαιτίας αυτού του κινδύνου υπάρχει πολύ ψηλό κόστος για αυτά. Αν είναι όμως έτσι, θα πρέπει να φροντίσουμε τα ποσά να χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά πλήρως. Να υπάρχει δηλαδή καλή απορρόφηση. Υπάρχει κάποιος έλεγχος για το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Θα μας βοηθούσε ίσως αυτό να βρούμε καλύτερες λύσεις στο μέλλον. Τώρα με τον κύριο Γκαλούσε και εκείνος το είπε ότι οργανώσεις που στηρίζουν τις επιχειρήσεις βρίσκονται σε χώδη κατάσταση. Και ίσως θα άξιζε τον κόπο να γίνει μια ταξινόμηση, να μπει κάποια τάξη σε αυτές. Και να υπάρχουν καλές προδιαγραφές για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνει αυτό, γιατί εύκολα το λέει κανείς. Να βάλουμε τάξη, ναι, αλλά έχουμε τον τρόπο, ξέρουμε πώς να το πετύχουμε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα παραδείγματα που ακούσαμε από το τελευταίο μιλητή. Εσείς είπατε ότι πρέπει να υπάρχει και ενθουσιασμός αλλά και λογική. Εσείς αναφέρατε πολλά καλά παραδείγματα και καλό θα ήταν να τα προωθήσουμε περισσότερο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μωράν τώρα. Ελίζπεθ Μωράν. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι η σημερινή ακρόαση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε ειδικού που είναι πραγματικά ειδικοί στο θέμα και που μας προσφέρουν και ένα προβληματισμό, αλλά μας δίνουν και συγκεκριμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρωτοβουλία. Θέλω να ρωτήσω τους ειδικού το εξή. Λένε, μας εξήγησαν πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε στους πιο φτωχούς με μικροπιστώσεις. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν πώς χρησιμοποιούν οι πιο φτωχές γυναίκες ε, τα μέσα μικροχρηματοδότησης. Σε διεθνές επίπεδο ξέρουμε ότι είναι οι γυναίκες εκείνες που είναι κυρίως οι δικαιούχοι και ζητούν τις μικροπιστώσεις αυτές. Τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η Ελίζα Σρέντερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Είδα και εγώ ξεκάθαρα ότι το παράδειγμα της Ουγγαρίας μας δείχνει ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τον μηχανισμό μικροπιστώσεων. Με εκπλήσει όμως το γεγονός ότι με ένα μικρό πρόγραμμα δεν χρησιμοποιείται τις δυνατότητες που δίνει το κοινωνικό ταμείο είναι σημαντικό γιατί για μερικά πράγματα προβλέπονται δάνεια από το κοινωνικό ταμείο. Άλλες χώρες το χρησιμοποιούν. Γιατί όχι η Ουγγαρία. Διότι αυτά που έχετε στη διάθεσή σας είναι πολύ λίγα για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όμως εδώ και 7 χρόνια δίνει τέτοιες δυνατότητες. Με εκπλήσει λοιπόν που δεν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με εκπλήσει επίση που βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ αργά και ότι παρουσιάζονται πολλές δυσκολίε. Από τη μια υπάρχουν βέβαια τα συγκεκριμένα παραδείγματα, υπάρχουν αυτοί που δίνουν τις μικροπιστώσεις. Είπατε όμως ότι χάνονται και χρήματα. Πολλοί χάνουν χρήματα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θέλει να πάει πιο μακριά και να δει πώς μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα. Εσείς λοιπόν ρωτάω Πώς δουλεύετε. η ενδιάμεση φορείς, η ενδιάμεση χρηματοδοτική φορείς ε, επομίζονται και αυτοί τον κίνδυνο ή όχι. Ποιος επομίζεται τον κίνδυνο τελικά. Εφόσον από την αρχή λέμε ότι πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό εμπόριο, αντίθετα ότι πολλές φορές χάνονται χρήματα. Θέλω να ξέρω λοιπόν από εσά πώς ακριβώς γίνεται αυτό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πώς ε, δουλεύετε, συμφωνείτε πρώτα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν ξέρω για σίγουρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από όσο ξέρω, δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει τον κίνδυνο, ούτε να πληρώσει γι' αυτόν. Ποιος λοιπόν αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Ευχαριστώ. Η King Kong τώρα σε γίνεται πιο γρήγορα. Κοιτάξτε, μια που δεν έχουμε αρκετό χρόνο, Ξέρω ότι σημειώνουν τις ερωτήσεις σας οι εμπειρογνώμονες. Μήπως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έτσι θα υποφεληθούν και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ σήμερα. Κοιτάξτε γιατί το κάνουμε, να σας εξηγήσω. Γιατί έχουν ακυρωθεί πολλές πτήσεις, πολλά τρένα. Πολλοί ευρωβουλευτές λοιπόν θέλουν να τελειώσουμε στις 4 το απόγευμα, αν είναι δυνατόν, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στα, στις εκλογικές τους περιφέρειες. Καταλαβαίνετε ότι είναι έκτακτη η σημερινή κατάσταση, γι' αυτό το ζητάω. Υπάρχουν όμως κάποια σοβαρά θέματα που ίσως να θέλετε να συζητήσουμε, κάποια θεμελιώδη ζητήματα. Ναι, ευχαριστώ. Ε, εγώ έλαβα κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που είχα θέσει. Βέβαια, ορισμένα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Όμως η ακρόαση αυτή ήταν ε, αρκετά ενδιαφέρουσα. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι δεν πιστεύουμε ότι οι μηχανισμοί μικροχρηματοδότησης είναι πανάκια και μπορούν να λύσουν όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Ε, δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αλλά η παρουσίαση του κυρίου Λάκη μας έδειξε ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες ε, όπως η Ρωμά. Αλλά υπάρχει η παρεξήγηση ότι οι πόροι ε, στην Ανατολική Ευρώπη πήγαν στους Ρωμά. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια να γιοχετευτεί ένα τμήμα των πόρων στους Ρωμά γιατί είναι ευάλωτοι. Ε, θέλω επίσης να ενθαρρύνω τον διαχειριστικό οργανισμό να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτές ε, τις μειονεκτούσες ομάδες. Είναι δυνατό κάτι τέτοιο και επίσης ε, θέλω να τονίσω κάτι που υπόθηκε νωρίτερα ότι η βασική υπόθεση είναι ότι το ESF θα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρηματοδοτήσει το κόστος ε, λειτουργίας και καθοδήγησης αυτών των οργανισμών. Αυτό είναι ουσιαστικό θέμα, ε, όμως ε, εδώ πρέπει να μιλάμε για ε, διασφαλισμένους πόρους η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν ε, ε, θέλει να στείλει κονδύλια αν δεν φτάνουν ε, αυτά τα κονδύλια στις μη ευάλωτες ομάδες και επίσης αναφερθήκατε στο ότι δεν είναι ρεαλιστικό να έχουμε 2% επιτόκιο όμως κοιτάξτε από το 2% μέχρι το 75% υπάρχουν και πολλά άλλα νούμερα και το να υπάρχει ένα επιτόκιο υψηλό ε, είναι αποδεκτό να έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε και την άλλη πτυχή. Θέλω να δω την πρώτη έκθεση και εγώ εμπιστεύομαι όσο είπατε ότι κάνετε προσπάθειες ε, να προσπαθήσετε να βρείτε ενδιάμεσους σε διάφορες χώρες. Αναφερθήκατε ε, σε αυτό το θέμα. Και θέλω να υποστηρίξω και όσο είπε και η Ελίζα ότι και για μένα ε, φαίνεται ότι προχωρά πάρα πολύ αργά η διαδικασία. Χρειάζεται χρόνο, στο ξέρω, χρειαζόμαστε και ένα πρόγραμμα επιχειρησιακό που να βοηθάει του ανθρώπου επί και να υπάρχουν και τα απαραίτητα στοιχεία ε, με τη χρηματοδότηση από το ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να έχουμε συνδυασμό και από αυτό το Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτός είναι ένας καλός συνδυασμός προκειμένου να συστήσουμε ένα πρόγραμμα που να λειτουργεί σωστά. Σας ευχαριστώ και περιμένω να δω την πρώτη έκθεση που θα είναι πιο ισορροπημένη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ε, την εισηγήτρια για τους Ρώμα ε, που είναι η επί της... Ε, έχουμε την έκθεση αυτή και η επόμενή μας συζήτηση είναι για τους Ρώμα. Ήθελα λοιπόν χρόνο για να ακούσουμε τη σχετική συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες. Ξέρω ότι όλοι κρατήσατε σημειώσεις. Εάν μπορείτε παρακαλώ να στείλετε email στην γραμματεία θα ε, μεταφέρουμε τις απαντήσεις σας όχι μόνο στους βουλευτές που έθεσαν τις ερωτήσεις, ε, αλλά με την άδειά σας θα διανύμουμε τις απαντήσεις σας και στους βουλευτές που δεν μπόρεσαν να παραβρίσκονται λόγω καιρού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι και αυτοί θα είχαν κάνει παρόμοιες ερωτήσεις αν θα μπορούσαν να έχουν έρθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μία τόσο δύσκολη μέρα με τόσο κακό καιρό. Ε, ελπίζω να μην έχετε δυσκολίες να επιστρέψετε. Πάντως άξιζε τον κόπο και ε, θα ήλπιζα να είχατε έρθει σε μία μέρα που να μην έχουμε τόσα προβλήματα με το χιόνι ε, σε τόσα κράτη-μέλη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Κίνγκα ε, Κόνης για να μας παρουσιάσει την έκθεση για τους Ρώμα. Κίνγκα, uh, um, uh, ε, τέσσερα λεπτά το πολύ. Θα δώσω τρία λεπτά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στους άλλους ομιλητές δύο λεπτά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, αν και υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις ανάμεσα στην ε, δημόσια κρόση μόλις ακούσαμε και ε, τα θέματα των Ρώμα, αν και δεν είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με το πλαίσιο και τις ε, συνθήκες. Ε, ξέρετε ότι η Επιτροπή μας είναι η συνδεδεμένη Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15. Ε, και η διάσκεψη των ε, Προέδρων έγινε αρκετά αργά, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να υποβάλω την έκθεσή μου πριν καν ε, ληφθεί η σχετική απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων και πριν καν έχουμε την τελική εκδοχή της επί της ουσίας αρμόδιας επιτροπής. Θα χρειαστούμε λοιπόν κάποιο χρόνο για τις λεπτομέρειες. Είχαμε χθε και προχθές μία δημόσια κρόαση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι το άλλο καθήκον μας θα είναι να συντονίσουμε το χρονοδιάγραμμά μας με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής. Υπάρχει μια σημαντική ημερομηνία. Η Κομισιόν είπε ότι θα υποβάλει την επόμενη ανακοίνωσή της που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης στις 9 Απριλίου και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την πρώτη εκδοχή της ανακοίνωσης της Κομισιόν πρωτού ε, εμείς οριστικοποιήσουμε τη δική μας έκθεση, διότι αλλιώς θα χάσουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε τα πράγματα και να συντονίσουμε τις εργασίες μας με αυτές τις επιτροπές. Επίσης, ε, επειδή αποτελεί προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία, θα συζητηθεί στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε λίγο περισσότερο πάνω στα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ε, χρονοδιάγραμμα. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη, δεν θα συζητήσω όλο το περιεχόμενο, διότι ε, έχετε την έκθεση αυτή και μάλιστα μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν ήθελα να πάρω τόσο πολύ... Δεν ήθελα να μιλάω στην γνωμοδότησή μου τόσο πολύ για ε, τα, τους βασικούς τομείς κοινωνικής ένταξης στο Ρώμα. Αυτό έχει καλυφθεί σε πολλές άλλες εκθέσεις. Ε, με ενδιαφέρει περισσότερο το πώς να εφαρμοστούν οι στόχοι αυτοί. Μιλώ για χρήση της ε, χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το πρόβλημα δεν είναι το ποσό της χρηματοδότησης, είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε στους ανθρώπους που πραγματικά ε, έχουν ανάγκη τα χρήματα αυτά. Ποιος θα πρέπει να υποφελείται, θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτος τύπος χρηματοδότησης και πιστεύω ότι πρέπει να ε, αναπτύξουμε περαιτέρω το σχετικό μέσο. Σημαντικό είναι στις εθνικές στρατηγικές για το 2020 να υπάρχει κεφάλαιο για την μείωση της στόχιας συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου για τους Ρώμα και τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους. Χρειαζόμαστε δεδομένα με βάση τις οδηγίες για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την χρήση των πόρων και σημαντικό είναι να ζητήσουμε και από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΣΑ, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας κλπ. να έχουν στις δικές τους εκθέσεις κεφάλαιο σχετικά με την κατάσταση στο Ρώμα. Θέλουμε ερεσιμότητα όσον αφορά ε, τα διαφορετικά ταμεία, θέλουμε mainstreaming, θέλουμε πολύ αυστηρή παρακολούθηση με βάση δείκτες ε, και benchmarks, μια αναφορά δηλαδή θέλουμε να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων Ευρωπαϊκών Ταμείων και συγχρηματοδότηση. Θέλουμε συντονισμένες δράσεις σε διάφορα επίπεδα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θέλουμε να καλέσουμε τις ε, εθνικές αρχές ε, να ε, συμμετέχουν στον προγραμματισμό, όπως επίσης και τους Ρώμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πολύ ευχαρίστως θα δω τις τροπολογίες σας και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες ώστε να έχουμε μια συνολική ε, έκθεση η οποία να μπορέσει να επηρεάσει τις εργασίες στο Συμβούλιο και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Κομισιόν που είναι ο σύμμαχός μας στο θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις τόσο λίγο όταν είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα. Να στραφώ αμέσως στην εισηγήτρια από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ και εγώ στην εκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα όμως να ευχαριστήσω την συνεισηγήτρια και σκιώδη Κιν Kong για την δικιά της γνωμοδότηση. Τα περισσότερα από τα θέματα που αναφέρετε στη γνωμοδότησή σας, όλα θα έλεγα, ταιριάζουν απόλυτα με την έκθεσή μου, οπότε τα υποστηρίζω απόλυτα. Επιτρέψτε μου όμως, αν μου επιτρέπετε, να έρθω λιγάκι και να σχολιάσω ορισμένα από τα σημεία που θίγεται. Το πρώτο και πιο σημαντικό όφελος από την γνωμοδότησή σας είναι όντως τα ταμεία. Και στην παράγραφο που ζητάτε να είναι πιο στοχοθετημένα, πιο ευέλικτα τα προγράμματα, μιλάτε και για συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα διάφορα ταμεία που πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των Ρώμα. Μιλάτε επίσης και για την αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση. Και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος για τις διάφορες οργανώσεις, μη κυβερνητικέ και άλλες που προσπαθούν να έχουν χρηματοδότηση για τους Ρώμα. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και τα υποστηρίζω απόλυτα. Ιδιαίτερα την βιωσιμότητα, γιατί όντως χρειάζεται μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Τέτοιου είδους προγράμματα όμως ε, δημιουργούν συχνά προβλήματα. Το Equal, για παράδειγμα, είδαμε πως βγήκε από το Κοινωνικό Ταμείο 2007-2013. Αυτό ήταν μια μεγάλη απώλεια. Αναφέρεστε επίσης στο συντονισμό, λέτε ότι πρέπει πρέπει να βελτιωθεί μεταξύ των οργανώσεων. Νομίζω όμως ότι και μεταξύ των πολιτικών πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Μεταξύ της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ε, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι συμπληρωματικά πράγματα. Η γραφειοκρατία, όπως πολύ σωστά λέτε, πρέπει να απλοποιηθεί. Να αποτελεί μεγάλο βάρος. Και όλοι οι φραγμοί που τίθενται στα ταμεία πρέπει να έρθουν. Ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα. Στις παράγραφους 13 και 14 αναφέρεστε στη σημασία που έχουν οι έρευνες που γίνονται για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Ρώμα. Λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λιγότερο περίπλοκα προγράμματα. Στην παράγραφο 8, στη δικιά μου την έκθεση, ζητάω νέα κριτήρια για διάφορες περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την διεκίζουν κυρίως ε, η Ρώμα, ώστε να μπορέσουμε να στοχεύσουμε πολύ συγκεκριμένα. Η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ άσχημη και ο πληθυσμός δεν είναι μόνο φτωχός εκεί, αλλά επιπλέον είναι σε ένα φαύλο κύκλο ένδυας, σε ένα σπιράλ αν δεν το κάνουμε, ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα παραλύσει. Αυτές τις ε, τόσο μειονεκτικές περιοχές που ζουν οι Ρώμα πρέπει να τις ενισχύσουμε. Ορισμένοι λένε ότι κοστίζει πολλά χρήματα. Εγώ όμως λέω ότι είναι φτηνότερο από τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν αργότερα, από την επιδείνωση δηλαδή των προγραμμάτων. Στην και 11 χαίρομαι που στηρίζετε την ιδέα ότι είναι ευθύνη της Κομισιόν. Και που ζητάτε από τα κράτη-μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους για την κοινωνική ενσωμάτωση που είναι όπως και απάλληψη της φτώχειας στόχος της Ευρώπης 2020. Όμως και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει πλήρης επικάλυψη μεταξύ των δύο πρωτοβουλειών, μερικώς ναι. Οι στόχοι των δύο στρατηγικών επικαλύπτονται σε ένα βαθμό, αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία που αναφέρονται στην έκθεσή μου και γι' αυτό χρειάζεται μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή στρατηγική που θα ενισχύει την ενσωμάτωση των Ρώμων. Τελευταία μου παρατήρηση Πάλι για την Κομισιόν. Να υπάρχει, ζητάτε, ένα ειδικό όργανο που θα ε, παρακολουθεί, θα παρατηρεί και θα αξιολογεί την δράση των χωρών για τους Ρώμα. Έξι χρόνια εδώ ζητάμε μια ειδική task force και όχι μόνο δύο ανθρώπους να δουλεύουν για τους Ρώμα κάπου. Όχι, θέλουμε κάτι υψηλότερο επίπεδο. Το Σεπτέμβριο άρχισε να υπάρχει αυτή η task force κάνει σοβαρή δουλειά, γιατί όντω παρατηρεί και διαπιστώνει που έχουν πάει τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Ρώμα. Αν ενισχυθεί, αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Έπειτα μιλάτε για δίκτες που θα βοηθήσουν να γίνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Το ζητάτε από την Επιτροπή αυτό, να φτιάξει αυτούς τους δείκτες ή από τα κράτη-μέλη. διότι εγώ πιστεύω πως η Επιτροπή, και αυτό θα υποστηρίξω στη Λίβη, ότι η Επιτροπή πρέπει να το κάνει αυτό, να φτιάξει δηλαδή ένα σώμα ειδικό που να κάνει αυτήν την αξιολόγηση με δείκτες από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί η διαδικασία θα είναι μια μακρά διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χίρς καταρχήν και κατόπιν η κυρία Ντελή. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρου ε, τη Σεσιλία που είναι σκιώδη συγγητρία. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το θέμα το Ρωμά είναι στην ατζέντα όλων των ε, σημαντικών ε, ε, θεσμών και ενδιαφερομένων. Πρέπει τώρα να εφαρμόσουμε όσο αποφασίσαμε και θεωρεί ότι η κυρία Γκόντς κάνει με την έκθεσή της ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση. Προτείνει να συμπεριλάβουμε τα εξή στη γνωμοδότηση. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κρατημέλη να έχουν ολιστική προσέγγιση όταν προσπαθούν να πετύχουν τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Πρέπει να τονίσουμε ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε τώρα είναι ότι ακόμη και η κατάσταση ε, βρίσκεται το θέμα των Ρωμά στην ημερήσια διάταξη. Είμαστε πολύ μακριά από τη λύση. Πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόσουμε όσα αποφασίσαμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται συντονισμό, πόροι και ενδυνάμωση των τοπικών αρχών και φορέων. Ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε είναι ότι πολλοί Ρωμά δεν έχουν ε, χαρτιά ε, και απλώς ε, μπορούν να τους αναγνωρίσουμε γιατί έχουν μείνει όλη τους τη ζωή στην ίδια χώρα τα κράτη-μέλη, στα κράτη-μέλη αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ε, το να μπορέσει κάποιο να αποδείξει ότι ανήκει σε αυτή την κοινωνία και στη χώρα, τον εμποδίζει να λειτουργεί στην κοινωνία. Πάρα πολλά παιδιά αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά. Ένα άλλο σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να γνωρίζουμε το παρελθόν μα. Ε, πρέπει να ε, διαδώσουμε πληροφορίε για την ιστορική κατάσταση στο Ρωμά Πρέπει να γνωρίσουμε τις εκθέσεις ε, της ε, Υπηρεσίας Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Η συνάδελφος θεωρεί ότι πρέπει να επενθυμίσουμε τις υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την επικότητα. Δεν μπορούν ε, να υπάρχουν διακρίσεις βάσει της φυλής του χρώματος της θρησκευτικής πεπίτης θρησκευτικών πεπιθήσεων κτλ. Επίσης πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι Ρωμά είναι Ευρωπαίοι πολίτες και όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχουν δικαίωμα όπως όλοι οι πολίτες ε, έχουν και αυτοί κοινωνικά και θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι το ένα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε για τους Ρωμά για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές. Ε, πρέπει να έχουμε πολιτικές με την ενεργή συμμετοχή των Ρωμά και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τους Ρωμά, κάτι αποφασιστικό σήμερα, γιατί ναι, η Ρώμα πάντοτε είναι αντικείμενο διακρίσεων, ε, ναι, ζουν σε άθλιες συνθήκες ε, και συχνά ζουν σε παράγκες, παραγκουπόλει. Ε, είναι απαράδεκτο η Ευρώπη για τη σε σχέση με τη μειονότητα αυτή να δίνει ε, τόσο κακή εικόνα, να αφήνει τον πληθυσμό αυτό σε τέτοια εξαθλίωση εδώ και αιώνε. Ήταν αντικείμενο διάκριση από τον υπόλοιπο πληθυσμό λόγω προκαταλήψεων. Σω θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και τον πολιτισμό των Αθήγανων, όπω και πολλού άλλου πολιτισμούς προωθούμε στη Γαλλία, γιατί όχι. Κάτι άλλο, κυρία Συγήτρια, ναι, πρέπει να στηριχθούμε στη χρηματοδότηση, αλλά ε, τι είναι η κοινωνική ένταξη, είναι η αναγνώριση των ε, ανθρωπινών αξιών. Πρέπει να έχουμε και μέτρα κοινωνικά, συνοδευτικά μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα. Ε, όταν ε, τους έχουν ε, δοθεί σπίτια, θα πρέπει να επιμείνουμε να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Θα πρέπει να τους προσφέρουμε πρόσβαση στις δημοσίες υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα. Είναι ουσιαστική ουσιώδες αυτό. Ε, επίσης για τις γυναίκες ε, που ανήκουν στη μειονότητα Ρωμά συνεχώς ε, είναι αντικείμενο διακρίσεων και το υπενθυμίσαμε αυτό. Η κυρία Χίρς το ξανά σήμερα το πρωί στην έκθεσή της. Υπάρχουν λοιπόν και σύνδεσμοι που πρέπει να υπενθυμίσουμε. Και τέλος, θέλω να επιμείνω στο ότι πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Περιφερειακό επίπεδο, τοπικό επίπεδο και οι αρχέ πρέπει να εμπλακούν. Είναι αναγκαιότητα αυτό και αληθεύει, αλλά πρέπει να κατευθυνθούμε και προ ε, μια διαπολιτιστική προσέγγιση, θα την αποκαλούσε εδώ, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ένταξη. Ευχαριστώ. Κυρία Μωρά. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου στις δύο συντάκτηρες των γνωμοδοτήσεων από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά και από τη δική μας Επιτροπή, αλλά και στη Λιβία Ρόκα, γιατί γνωρίζουν πραγματικά εις βάθος τα ζητήματα αυτά και νομίζω ότι εδώ Πρέπει να παραδεχτούμε ότι όσα γνωρίζουμε εμείς ε, περιορίζονται στα στερεότυπα και δεν έχουμε εις βάθος γνώση της κατάστασης. Ε, έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι εφόσον γνωρίζουν τόσο καλά το ζήτημα, ε, τις εμπιστεύομαι και δεν θέλω εδώ να κάνω δηλώσεις δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Καταρχήν, συμφωνώ με όσοι υποθήκαν για την στρατηγική πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πρώτη μας ενσυχία ότι δηλαδή τα ε, κορδίλια από τα διαφορετικά ταμεία για την ένταξη στο Ρωμά να κατορθώνουν να στηρίζουν τις πολιτικές ε, ένταξης ε, των Ρωμά είχαμε ε, κάποιες πληροφορίες ε, από την ε, αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τους την προηγούμενη φορά και μας έδειξε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή αποτελεσματικές στρατηγικές σχετικά με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο εγώ συμφωνώ με τη Λιβία Ροκά ότι ο πληθυσμός στο Ρωμά συνδέεται με περιφέρειες όπου δεν υπάρχει οικονομική δυναμική. Δηλαδή μιλάμε για μια κοινωνική φτώχεια περισσότερο παρά για μια περιφερειακή φτώχεια. Και επειδή είναι ριζωμένη η φτώχεια αυτή εκεί, μας κάνει να μπαίνουμε ε, σε ένα φαυλοκύκλο, σε ένα σπιράλ εγώ νομίζω ότι πρέπει ακριβώς να αφοσιωθούμε στο εξή να συγκλίνουμε πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές για να βγάλουμε τον πληθυσμό αυτό και τις συγκεκριμένες περιφέρειες από τη φτώχεια. Στην τελευταία μας επίσκεψη στην Ουγγαρία για την προετοιμασία της Ουγγρικής Προεδρίας Προέκυπτε πολύ συχνά μια τέτοια ανάλυση και νομίζω ότι από αυτού πρέπει να εργαστούμε. Το τρίτο σημείο αφορά τη μόχλευση, στο μοχλό της επανένταξης. Το πληθυσμό αυτών αναφέρεστε, κύριε Αγκόν, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στην απασχόληση. Αναρωτιέμαι το εξή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αναρωτιέμαι πώ θα έπρεπε να πάμε πιο μακριά. Ε, ό,τι αφορά την οικογενειακή ενότητα, έτσι ώστε και τα ίδια τα παιδιά να λαμβάνουν μια ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Δεν αρκεί, θεωρώ, η εκπαίδευση για αυτό το ρομαδικό πληθυσμό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια δουλειά σε σχέση με το ρόλο και την ευθύνη των γονέων απέναντι στα παιδιά. Θέλω να σας θέσω και μια ερώτηση που έχει να κάνει με το σημείο 6 την ε, υποχρεωτική θεσμική εγγύηση. Και θέλω να μου πείτε για ποια εγγύηση ακριβώς μιλάτε. Φυσικά πρέπει να αξιολογήσουμε τις πολιτικές, αλλά τι ακριβώς εννοείται όταν αναφέρεστε σε αυτήν την υποχρεωτική θεσμική εγγύηση. Θέλω πάντως ε, να ε, σας ευχαριστήσω και τις δύο για το έργο σας. Ευχαριστούμε. Η συγγήτρια Κόγκ, μήπως να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά, εντάξει. Ναι, μετά πρέπει να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Κόγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ουσιαστική συζήτηση που είχαμε. Λυπάμαι που είμαστε τόσο λίγοι, αλλά βέβαια νομίζω ότι πιο σημαντικοί ήμασταν εδώ. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις σας στην συγκήτρια. Ε, κοιτάξτε, προσπάθησα όντως να προσθέσω κάποια πράγματα που εσείς δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε στη δικιά σας έκθεση, γιατί εσείς εκπροσωπείτε τη ΛΥΒΕ. Αλλά πρέπει να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση, το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα θέματα διακρίσεων είναι εξίσου σημαντικά, το καταλαβαίνω. Ε, δεν τα έβαλα εγώ γιατί θεώρησα ότι εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με τα κοινωνικο-οικονομικά και εσείς ασχολείστε πιο πολύ με τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα προσπαθήσουμε στο τέλος να συμπεριλάβουμε και τα μεν και τα δε βέβαια. Οι δείκτε στα κριτήρια νομίζω ότι πρέπει να τεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω. Μπορούμε να το διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρα. Ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν benchmarks που να καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω επίση ότι η Task Force είναι καλό να είναι ως μόνιμη. Νόμιζα ότι ήταν προσωρινή μέχρι τώρα. Να γίνει μόνιμη. Να υπάρχει δηλαδή ένα σώμα το οποίο να δουλεύει πάνω σε αυτό, σε υψηλότερο επίπεδο. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Για τη Σεσίλια Βίλκστρομ που την ε, εκπροσωπείτε εδώ. Ελεύθερη διακίνηση είπα ότι θα καλυφθεί από τη ΛΥΜΠΕ. Για το συντονισμό και τους πόρους συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό και περισσότερο πόρους, αλλά σίγουρα περισσότερο ε, συνολική άποψη, σφαιρική συντονισμό. άρα. Για το θέμα της εδαφικότητας συμφωνώ ευθύς εξ αρχής. Είναι ένα μέρος του προβλήματος γιατί όντως τα προβλήματα συγκεντρώνονται σε έναν χώρο πολλές φορές. Άρα συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση η Ουγγαρία έχει προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για να καλύψει τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τις πιο μειονεκτικές βέβαια που έχουν λιγότερο σε σχέση με το ΕΠ κλπ και νομίζω ότι μπορούμε αυτή την προσέγγιση να την χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα σε αυτές τις μικρές περιοχές πολλές φορές δεν υπάρχουν καν κοινοφελείς υπηρεσίες. Και αυτό να το πούμε. Τα παιδιά φυσικά και είναι στο επίκεντρο του θέματος. Η εκπαίδευση, τα σχολεία, ε, τα παιδιά να πηγαίνουν ε, σχολείο από τη μικρή ηλικία, ναι, Τώρα με ρωτήσατε να σας πω τη γνώμη μου για την αρισιμότητα. και για την ε, απάλληψη των διακρίσεων, της γετοποίησης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνεισφέρουν στην ε, απάλληψη των ε, διακρίσεων. Δεν βελτιώνουν ε, την κατάσταση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να υπάρξει μια αποκατάσταση. Δηλαδή σε μια πόλη, σε ένα μέρος, να μην καταλήγουν να αποκλείονται από μια περιοχή η οποία επιδεινώνεται και να καταλήγουν σε γκέτο. Αντίθετα πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωσή τους. Αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε ως προσέγγιση. Κατά τα άλλα, δεν ε, θέλω να καθυστερήσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τις τροπολογίες σας θα δουλέψω φυσικά και με τους Κιώδης και με τη Λίβια και θα φροντίσουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση που να περιλαμβάνει και την γνωμοδότησή μας. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ θα είχα να κάνω κάποιε παρατήρησει, αλλά δεν πειράζει, θα τι πω αργότερα στην εισηγήτρια. Η... Με τι τροπολογίε. Θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε. Προθεσμία είναι Δεκεμβρίου. 24 Ιανουαρίου θα δούμε εδώ τι τροπολογίε και θα ψηφίσουμε στις 25 Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσουμε με την κοινή συζήτηση όσον αφορά τον προπολογισμό και την απαλλαγή. Οι συντονιστές έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή αυτή που έχουμε κάνει στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω ότι εφόσον όλα πάνε καλά, τέσσερις η ώρα να έχουμε τελειώσει. Και έτσι θα μπορέσετε όλοι να επιστρέψετε Φαντάζομαι ότι το θέλετε και εσείς και διερμηνείς λέει η Πρόεδρος. Ελπίζω 4 ώρα να έχουμε τελειώσει τις εργασίες μας σήμερα το απόγευμα.